Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, θα σα πρότεινα να αρχίσουμε τι εργασίε μα. Σα παρακαλώ λίγη ησυχία. Είδατε την ημερήσια διάταξή μα και αν δεν έχετε σχόλια θα θεωρηθεί εγκεκριμένη. Σήμερα το απόγευμα θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους ε, των Γκένσε και Τζέσε και καλωσορίζω τις παρούσες προσωπικότητες. Θα επανέλθω στη συνέχεια στην παρουσίασή τους. Αύριο το πρωί θα έχουμε και πάλι ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους της Ανδόρα, Λίχτενστόιν και Μονακό και αύριο το απόγευμα από τις 3 μέχρι τις 6.30 ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους τεσσάρων πολυεθνικών εταιριών που τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα της Επιτροπής μας τα θέματα που μας απασχολούν και μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ανακοινώσεις του Προέδρου, σας επιβεβαιώ ότι έχουμε όλες τις γλώσσες εργασίας της Επιτροπής μας, δεδομένων των αναγκών των μελών. Έχουμε λοιπόν διερμηνία σε όλες τις γλώσσες και ευχαριστώ τους διερμηνείς. Ευχαριστούμε. Και όπως σε όλες μας τις συνεδριάσεις και η παρούσα είναι δημόσια, δηλαδή είναι ανοιχτή για το κοινό, για, το κοινό, για τον τύπο και μεταδίδεται και απευθείας ε, στο διαδίκτυο με web streaming. Στο σημείο 3, έγκριση των πρακτικών. Τη περασμένης συνεδρίασης, αν δεν έχετε καμιά αντίδραση μέχρι το τέλος της συνεδρίασης σήμερα, θα θεωρηθούν εγκεκριμένα και τα πρακτικά τις περασμένης συνεδρίες, 29 Φεβρουαρίου 2016. Περνάμε λοιπόν αμέσως στην ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους των Ίσον Γκένσλε και Τζέρσι. Με χαρά καλωσορίζω τον κύριο Ρομπ Γκρέι που είναι Διευθυντής Διεθνούς Φορολογίας του Γκένζεϊ και τον κύριο Colin Powell, mm. που είναι ε, σύμβουλος του Chief Minister του Γκένζεϊ για τις διεθνεί υποθέσεις. Είχα άλλωστε την ευκαιρία όσο και την τιμή να τον ε, δεχτώ, ε, τον Πρωθυπουργό συγκεκριμένα Γκένζεϊ και Τζέρζεϊ, στο περιθώριο της προηγούμενης Επιτροπής ΤΑΞ 1. Πριν μας παρουσιάσουν τη φορολογική κατάσταση οι προσκεκλημένοι στο Γκένσε και Τζέρσι και κατόπιν αιτήματο των συντονιστών προσκάλεσα τον κύριο Μουταρδιέ, Γενικό Διευθυντή της Ταξιούντα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας κάνει μια παρουσίαση της κατάστασης αυτών των δικαιοδοσιών καθώς επίσης και τις σχέσεις με το εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι τμήμα του προγράμματος που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο. Θα παρακαλώ τον κύριο Μουταχλιέ λοιπόν να μας κάνει μια παρουσίαση οκτάλεπτη το πολύ περίπου και μετά θα ακούσουμε τους προσκεκλημένους από τον Γκέρνζα και τον Τσέστε και θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και απαντήσεις με τα μέλη και τους εισηγητές μας. Κύριε Διευθυντά, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Με ιδιαίτερη χαρά έρχομαι να δούμε πώς έχει η κατάσταση ε, σε σχέση με αυτές τις χώρες τις οποίες ακούσετε και εσείς ε, Γένσε, Τζέρσε, Λίχτενστάιν, Ανδόρα και Μονακό έχουμε συνεργασία μαζί τους είναι ευρωπαϊκές δικαιοδοσίες πλην ε, όχι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, των εταιριών έχουμε ένα νέο διάλογο με κάθε μία από τις χώρες. Ξέρετε ότι οι σχέσεις μας οι θεσμικές δεν είναι ομοιογενείς ούτε τα διάφορα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και στις συζητήσεις μας με αυτές τις ε, δικαιοδοσίες αλλά τα θέματα που μας απασχολούν στη συνεργασία μας είναι τα ίδια. Πρόκειται λοιπόν για βελτίωση της φορολογικής διαφάνειας, της σχέσης που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη και οι πέντε αυτές δικαιοδοσίες, αλλά και θα πρέπει να συζητήσουμε και άλλα θέματα φορολογικού αθέμητου ανταγωνισμού, ιδιαίτερα ε, στα πλαίσια του κώδικα δεοντολογίας για την φορολόγηση των επιχειρήσεων. Αν μου επιτρέπετε θα πω δύο λόγια για το πώς έχει σήμερα η κατάσταση και θα καταλήξω ε, με τις μέλουσες εξελίξεις, ε, πώς τις βλέπουμε και πώς βλέπουμε να διαγράφονται και να διαμορφώνονται οι σχέσεις μας με τις χώρες αυτές. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση των σημερινών θεμάτων, επιτρέψτε μου να αρχίσω από το ζήτημα της φορολογικής διαφάνειας. Έχουμε ενισχυμένο διάλογο εδώ και μια δεκαετία ε, με το σύνολο των χωρών αυτών και τις πέντε χώρες δηλαδή, διαφορετικό από χώρα σε χώρα με το Λίχτενστάιν, την Ανδόρα, το Μονακό, τον Άγιο Μαρίνο και την Ελβετία σε ό,τι αφορά τη φορολογική διαφάνεια έχουμε διμερείς ε, συμφωνίες. Ε, το ένα μέρος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το άλλο συμβαλόμενο είναι η κάστοτε χώρα. Σε ό,τι αφορά τώρα τα εδάφη που ε, συνδέονται και εξαρτώνται από τις κάτω χώρες και ε, το Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι η περίπτωση του Γκέρζε και του Τζέρσεϊ, έχουμε ένα γενικό κοινοτικό πλαίσιο το οποίο υλοποιείται μέσω διμερών συμφωνιών μεταξύ των κρατών μελών πλέον και αυτών των ε, επικρατιών, των εδαφών που συνδέονται ή εξαρτώνται από τις κάτω χώρες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πώς εξασφαλίζουμε τώρα τη φορολογική διαφάνεια. Όλες αυτές οι χώρες και οι δικαιοδοσίες έχουν ακολουθήσει το δρόμο της φορολογικής διαφάνειας με αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τα τραπεζικά δεδομένα ε, το 2013-2014 ε, θα ακούσετε σήμερα τι γίνεται στο Γκένζεϊ και στο Τζένζεϊ, αλλά και στο Λίχτενστάιν και στο Σαν Μαρίνο αργότερα τι έχουμε κάνει εκεί ε, υπάρχει αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και μάλιστα ταχεία διότι από φέτος έχει αλλάξει το σύστημα, δεν είναι κατόπιν αιτήματο, είναι αυτόματη η ανταλλαγή πληροφοριών, ενώ άλλε δικαιοδοσίε όπω είναι η Ανδόρα, Μονακό αλλά και η Ελβετία θα ε, υιοθετήσουν τις νέες προδιαγραφές αυτές το 2017. Όπως γνωρίζετε, οι διμερείς συμφωνίες τις οποίες έχουμε συνάψει με την Ελβετία, το Λίχτεστάιν, την Ανδόρα, το Μονακό και το Άγιο Μαρίνο έχουν ε, ανανεωθεί και ήδη ισχύουν ορισμένες, ενώ άλλες ε, είναι στο στάδιο της ολοκλήρωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συμμετάσχει πλήρως σε αυτές τις εργασίες που επιτρέπουν να διευρυνθεί το σύστημα που έχουμε εμείς τα 28 κράτη-μέλη τώρα και να επεκταθεί προς τις δικαιοδοσίες αυτές. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Γκένζε και το Τζέζι, οι σημερινές ε, συμφωνίες έχουν περάσει, όπως σας είπα, από την ε, ανταλλαγή ε, κατόπιν αιτήματος στην αυτόματη, έχουν αναπροσαρμοστεί οι συμφωνίες και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτή η μετάβαση είναι αντικείμενο συνεχούς και διαρκούς διαλόγου με τα κράτη-μέλη σε ένα επίπεδο υψηλό, σε μια ομάδα υψηλού επίπεδου για τη φορολογία έτσι ώστε οι νέες ε, συμφωνίες να υλοποιούνται με τρόπο συντονισμένο και αποτελεσματικό. Δύο λόγια τώρα για θέματα θέμη του φορολογικού ανταγωνισμού. Όπως γνωρίζετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει κώδικα δεοντολογίας για την φορολόγηση των επιχειρήσεων που είναι καθοδόν. Σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική τώρα φιλοδοξία που έχουμε είναι να καλύψει όσο γίνεται περισσότερες χώρες. Από την αρχή των εργασιών για τον κώδικα διοντολογίας, το σύνολο των κρατών ε, και των εδαφών που εξαρτώνται από τις χώρες μας και το Γκένζε και το Τζέσι συμμετείχαν πλήρως σε αυτό τον κώδικα. Δηλαδή αυτές οι δικαιοδοσίες καλύπτονται, εξετάστηκαν ως προς το συμβατό των συστημάτων τους για το φόρο των επιχειρήσεων πάντα, σε σχέση με κριτήρια της ε, χρηστής ε, φορολογικής διαχείρισης, ήδη από την αρχή των εργασιών. Και κάθε φορά που θεωρήθηκε αυτό απαραίτητο, ε, όταν η ε, χώρια νομοθεσία κάστοτε ήταν υπό αναθεώρηση. Για τις τρίτες τώρα χώρες διαφέρει η κατάσταση. Το 2013 και 2014 είχαμε ένα ειδικό διάλογο με την Ελβετία, που κατέληξε στην υπογραφή ενός μνημονίου κατανόησης έτσι ώστε να καταργηθούν κάποια συστήματα φορολογίας επιχειρήσεων που είτε σε ε, συνομοσπονδιακό ελβετικό επίπεδο είτε σε επίπεδο καντονιών. Ε, ίδιο διάλογο έχουμε αυτό το καιρό με το Λίχτενστάιν και μετά την ολοκλήρωσή του ορισμένα φορολογικά καθεστώτα πάντα ε, για τις επιχειρήσεις στο Λίχτενστάιν θα εξεταστούν στα κράτη-μέλη στα πλαίσια αυτού του διαλόγου. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ειδικό διάλογος ε, με άλλες χώρες όπως είναι η Ανδόρα, το Μονακό ή ο Άγιος Μαρίνος. Ιδού λοιπόν με δύο λόγια ε, το πού βρίσκεται ο διάλογος για τη φορολογική διαφάνεια και πώς εξετάζουμε τα φορολογικά καθεστώτα που ενδεχομένως να είναι επιζήμια ή να έρχονται σε σύγκρουση ε, στις δικαιοδοσίες τις οποίες θα εξετάσετε σήμερα και αύριο. Να πω δύο λόγια ακόμα για το τι μέλη γενέστε, πώς βλέπουμε ε, τη συνέχεια των εργασιών. Θα πρέπει να υλοποιηθεί μια εξωτερική στρατηγική που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Ιανουάριο είναι ένα από τα στοιχεία του πακέτου για την καταπολέμηση της ε, φορολογικής βελτιστοποίησης, όπως ονομάζεται. Όπως ξέρετε, έχουμε ε, εντοπίσει μια διαδικασία σε τρία στάδια για να ε, ελέγξουμε και να εξετάσουμε τι κάνουν κάποιες τρίτες δικαιοδοσίες έτσι ώστε να έχουμε ένα σύστημα με λίστες πανευρωπαϊκές κρατών που δεν συνεργάζονται, που είναι μη συνεργάσιμα. Σας είπα λοιπόν τρεις φάσεις, τρία στάδια. Το πρώτο θα αρχίσει και θα είναι μια ανάλυση ε, της κατάστασης στις τρίτες χώρες ε, σε σχέση με το πώς εφαρμόζουν ε, τα κριτήρια της χρηστής διαχείρισης ε, και με αντικειμενικό τρόπο και με αντικειμενικά κριτήρια για να έχουμε ανάλυση κινδύνου ε, δεδομένων των ειδικών οικονομικών ε, σχέσεων που έχει Ένωση με τις δικαιοδοσίες αυτές. Αυτό το πρώτο στάδιο αναμένεται να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο. Στη συνέχεια θέλουμε να έχουμε συζήτηση με τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να εξετάσουμε ποιες είναι εκείνες οι δικαιοδοσίες με τις οποίες θα πρέπει κατά προτεραιότητα να προχωρήσουμε σε ένα διάλογο για να εξετάσουμε εάν και πώς εφαρμόζονται αυτά τα κριτήρια. Και αφού τελειώσει αυτός ο διάλογος και σε περίπτωση που δεν αποδειχθούν συνεργάσιμες κάποιες δικαιοδοσίες, τότε και μόνο τότε θα ε, συνταχθεί ένας πανευρωπαϊκός κατάλογος. Ε, θα μπορούσε να αλλάξει λοιπόν το είδος ε, του διαλόγου ε, που έχουμε με τρίτες χώρες. Δεύτερο στοιχείο. Ο κώδικα διοντολογία ο ίδιο εξελίσσεται διότι τα κράτη-μέλη αναθεωρούν την εντολή του. είναι δυνατό και πιθανό να χρειαστεί να επανέλθουμε στι χώρε αυτέ και να δούμε πώ μπορεί να επηρεάσει αυτό το διάλογο μα μαζί του στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται ο κώδικα διοντολογία. Τελευταίο και θα κλείσω με αυτό βελτιώσαμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία για κάποια σημεία πολύ σημαντικά όπως είναι αυτόματη ε, ανταλλαγή των tax rulings ή την έκθεση αναχώρα, country by country reporting, ε, να λέει κάθε εταιρεία δηλαδή που έχει ποια κέρδη σε ποια χώρα. Τα ίδια αυτά στάνταρ, ίδιες προδιαγραφές θα δούμε και θα πρέπει να εφαρμόζονται και από τις ευρωπαϊκές δικαιοδοσίες από κράτη που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δούμε πώς τα κράτη-μέλη θέλουν να παρακολουθούμε την ε, χρηστή και σωστή υλοποίηση όλων αυτών. Ελπίζω αυτή η επισκόπηση ήταν αρκετά ε, λεπτομερής και εμπεριστατωμένη για να σας βοηθήσει ε, στη συζήτηση που θα έχετε με τις αλόγω λόγω δικαιοδοσίες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά για αυτή την εικόνα που μας παρουσιάσετε στο θέση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρουσιάσετε τις σχέσεις νομικές και πολιτικές με τις δικαιοδοσίες που θα ακούσουμε σήμερα και, και αύριο. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ρόμπ Γκρέι εν ονόματι του Γκέντζε. Λοιπόν, κύριε Διευθύντα, περίπου 8 λεπτά έχετε στη διάθεσή σας για να μας ενημερώσετε. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αξιότιμοι βουλευτές της Επιτροπής Tax ε, 2. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι σήμερα εδώ ε, για να ανταλλάξουμε απόψει. Λέγομαι Ρομπ Κρέι και όπω είπε ο πρόεδρο, ε, είμαι διευθυντή τη Διεθνού Φορολογικής Πολιτική τη κυβέρνηση του Γκένση και μέχρι το τέλο του 2015 ήμουν διευθυντή του Φόρου Εισοδήματος. Θα είμαι σχετικά σύντομος στην εισαγωγική μου παρέμβαση, διότι έχετε λάβει ήδη πολλές από τις λεπτομέρειε στις επιστολές ε, των Προέδρων των τοπικών κυβερνήσεων του Γκουένση και Τζέρσι με ημερομηνία 22 Φεβρουαρίου 2016, καθώ ε, και στις ε, αναλυτικές, στα αναλυτικά κείμενα που εστάλησαν σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις tax rulings το Μάιο του 2015. Η Γραμματεία επίση θα σα διανύμει ένα κείμενο με κάποια στοιχεία τα οποία θα παραλείψω στην εισαγωγή μου για να είμαι σύντομο. Από την αρχή η κυβέρνηση του Γκουένση ε, ψήφισε ομόφωνα να ε, παραμείνει δεσμευμένο ε, να εφαρμόσει τα διεθνή πρότυπα. Και αυτό δεν αποτελεί επιλογή για μας, αποτελεί ευθύνη. Εγώ εκπροσωπώ τον Γκουένση την ομάδα εργασίας του ΟΣΑ για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και στην ομάδα ad hoc BEPS για το πολυμερές μέσο και Επίσης ε, το Γκέρνσι θα είναι πλήρες ε, μέλος ε, του Διεθνούς Φόρουμ και παίρνουμε πολύ στα σοβαρά τα πράγματα αυτά, κάτι που φαίνεται από το γεγονός ότι δημιουργήθηκε το, το Παγκόσμιο Φόρουμ μάλλον ε, κατόπιν πρόταση του Γκέρντσι αποφασίστηκε ε, να πραγματοποιείται τη ε, συνάντηση για των αρμοδίων αρχών. Το Γκέρντσι αποτελεί εξαρτώμενο έδαφο του Ηνωμένου Βασιλείου όπω και το Τζέρσι. Αυτό είναι τελείω διαφορετικό καθεστώ από το καθεστώ των υπερπόντιων εδαφών όπω είναι το Γιβραλτάρι ή η Παρθένη νήση. Το Γενση δεν εκπροσωπείται στο Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου και δεν αποτελεί μέρο του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου δεν νομοθετεί για τον Γκέντσι χωρί τη συγκατάθεσή του. Ενώ συνταγματική πρακτική είναι το Ηνωμένο Βασίλειο να συμβουλεύεται τον Γενση προτού να το δεσμεύσει στο διεθνέ δίκαιο κατόπιν συμφωνία των Γκένση έχει ε, συμπεριληφθεί σε διάφορε διεθνεί συμβάσει που έχει προσυπογράψει το Ηνωμένο Βασίλειο. Για παράδειγμα, το 1991 η σύμβαση του ΩΣΑ αποφασίστηκε να καλύπτει και τον Γκένση ε, κατόπιν αίτηση του Γκένση. Και έτσι ισχύουν οι αποφάσει και οι συστάσει του ΩΣΑ με τον ίδιο τρόπο για τον Γκένση όπω και για το Ηνωμένο Βασίλειο. Η σχέση του Γκένση με το Ηνωμένο Βασίλειο προβλέπεται από το πρωτόκολλο 3 της, ε, σύμβασης προσχώρησης, ε, συνθήκης προσχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα το 1972, σύμφωνα με ε, την οποία το Γκέρνσι αποτελεί μέρος του τελωνιακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει ελεύθερη διακίνηση ακαθών μεταξύ του Γκέρνσι και των κρατών μελών. Το Γκέρνσι ωστόσο δεν αποτελεί μέρος της ενιαίας αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και δεν απαιτείται να εφαρμόζει τις σχετικές οδηγίες. Επίσης, αποτελεί τρίτη χώρα όσον αφορά την φορολογική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο μπορούμε ε, οικειοθελώς να εφαρμόζουμε κάποια μέτρα όπως ε, συνέβη με την ε, οδηγία για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων. εφαρμόζουμε όλες, ε, όλα τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών ώστε να μην αποτελούμε ε, κρυφή λύση για να ε, μεταβιβάσει κανεί σε συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία. Έχουμε καθεστώς φορολογικό το οποίο πληρεί τα πρότυπα του ΩΣΑ όσον αφορά τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών. Ο ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματο είναι 20%. Υπάρχει γενικό κανόνα ε, για την φοροαποφυγή και η φορολογική απάτη αποτελεί αδίκημα και στον Κέρνση. Οι επιχειρήσεις ε, γενικά ε, πληρώνουν μηδενικό φόρο, ωστόσο κάποιες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες φορολογούνται με 10% ενώ επιχειρήσεις κοινή ωφελία και επιχειρήσεις που λαμβάνουν τόκους ε, από εδάφη στο ε, φορολογούνται με 20%. Επίσης, το, φορολογικό, ε, το εταιρικό φορολογικό καθεστώς ε, συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και είναι ένα σύστημα το οποίο προστατεύει την οικονομία του νησιού και διασφαλίζει την φορολογική ουδετερότητα ο φορολογικός εταιρικός συντελεστής ε, του 0% βασίζεται ε, στην ε, αρχή της μη διάκρισης της ομάδας του κώδικα διοντολογίας. Ως Διεθνές Κέντρο Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών συγκεντρώνουμε κεφάλαιο, διευκολύνουμε την επένδυση στις ευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές αγορές. Ε, τα έσοδα των επενδυτών θα πρέπει να φορολογούνται στην πατρίδα τους ε, και οι σχετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες ε, θα πρέπει να φορολογούνται στον τόπο που πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες αυτές, κάτι που ευθυγραμμίζεται με το θεματολόγιο BEPS για την μεταβίβαση κερδών και τη συρρήκνωση της φορολογικής βάσης. Το Γκένσι δεν είχε φορολογικές αποφάσεις τύπου tax rulings από το 2008. Ε, ε, Τότε που εισήχθη δηλαδή το ε, ισχύον καθεστώς εταιρικής φορολογίας. Ενώ οποιασδήποτε αποκλήσεις από την νομοθεσία αντιμετωπίζονται με δηλώσεις πρακτικής statements of practice. Επίσης, ε, δεσμευτήκαμε να συμμετάσχουμε στην πρωτοβουλία του ΟΣΑ για την διαφάνεια και την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών το 2002. Για παράδειγμα, ε, συμμορφωνόμαστε με τις αρχές του κώδικα διοντολογίας για την ε, εταιρική φορολογία. Και το σύστημά μας Επίσημώ εγκρίθηκε από την ε, ομάδα δεοντολογίας το Δεκέμβριο του 2012. Επίσης, ε, οικειοθελώ ε, εφαρμόσαμε την οδηγία για τη φορολογία των αποταμιεύσεων. Συμμετέχουμε επίσης στην ομάδα των πρώτων που υιοθέτησαν τα κοινά πρότυπα υποβολή εκθέσεων. Έγινε αξιολόγηση από το Παγκόσμιο Φόρουμ του ΟΣΑ όσον αφορά την διαφάνεια και θεωρήθηκε ότι συμμορφωνόμαστε με τα διεθνή πρότυπα για την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αίτηση. Ε, έχουμε δηλαδή την ίδια βαθμολογία στο σημείο αυτό με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τι Ηνωμένε Πολιτείε και άλλου. Συμμετέχουμε στην ε, πολιετή ε, σύμβαση για την ε, αμοιβαία διοικητική αρρωγή και επίσης σύντα διμερείς συμφωνίες ε, για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών συμπεριλαμβανομένων 23 με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 13 διμερείς συμφωνίες διπλής φορολογίας επικροτούμε την ε, θετική αυτή αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τον ΩΣΑ. Το Γκένσι όπως και το Τζέρσι ε, πληρεί τα διεθνή πρότυπα για την φορολογική διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών και οι πολιτικοί μας έχουν καταστήσει σαφές ότι θα συνεχίσουν να το κάνουν αυτό με ομόφωνη πολιτική απόφαση. Τα επόμενα βήματα ε, συμμετέχουμε ενεργά όσον αφορά το θεματολόγιο BEPS. Και το Γκένσι και το Τζέσι συμμετέχουν στην ομάδα ad hoc BEPS για το πολιετές μέσο και το Γκένσι στηρίζει τις δράσεις για να διασφαλιστεί ε, ότι το διεθνές σύστημα είναι δίκαιο. Το Γκένσι δεν έχει ε, εκτενές δίκτυο συμφωνιών διπλής φορολογίας και γι' αυτό δεν χρησιμοποιείται για τη μεταβίβαση κερδών και για τις ε, τιμές μεταβίβασης. Ωστόσο, είναι σημαντικό παρόλα αυτά να παίζουμε ενεργό ρόλο στην εφαρμογή των διεθνών αυτών προτύπων, κάτι που ταιριάζει με την προσέγγισή μας να φροντίσουμε ο χρηματοπιστωτικός μας ε, τομέας να έχει πραγματική ουσία. Επικροτούμε τα βήματα που έχουν γίνει όσον αφορά το benchmarking και την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών για την αντιμετώπιση της ε, επιθετικής ε, φορολογικής ε, απάτης και σχεδιασμού. Σύντομα, οι υπουργοί μα ε, θα συστήσουν στο Κοινοβούλιο τον Κέρνση να υιοθετήσει και την υποβολή εκθέσεων αναχώρα. Όσον αφορά το θέμα τη πραγματική ιδιοκτησία, ε, τον Κέρνση είχε ένα αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο ε, για τις εταιρείε καταπιστευμάτων και επίσης συμμεριζόμαστε τον στόχο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά ε, την έγκαιρη ε, ανταλλαγή πληροφοριών για την πραγματική κυριότητα. Στόχος μας είναι στον Γκένσι να έχουμε ασφαλές μητρό όπου να αναφέρεται και το σημείο επαφής. Έχουν ξεκινήσει εργασίες και το 2017 θα υποβληθούν ε, προτάσεις στο Κοινοβούλιο προς έγκριση. Έτσι κλείνω την ε, εισαγωγική μου παρέμβαση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Κόλιν Πάουελ, εν ονόματι του Τζέρσι έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ Προέδρε, δικαιωμένα μέλη της Επιτροπής ΤΑΞ 2. Να σας παρουσιαστώ είμαι ο Κόλιν Πάουλ και είμαι σύμβουλος του Υπουργού της Κυβερνήσεως για Διεθνείς Υποθέσεις κυρίως για διεθνείς πρωτοβουλίες για φόρους, χρηματοοικονομικούς κανονισμούς και καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος. Εκπροσωπώ την κυβέρνηση ε, του Τζέρσι και χαίρομαι που μπορώ να συναντηθώ με την Επιτροπή σας. Και εμείς θεωρούμε ότι απαιτείται διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις αρχές της φορολογικές και επιβολής του νόμου σε σφαιρικό επίπεδο η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Συμφωνούμε ότι αυτοί που δεν συμμορφώνονται με τις διεθνείς προδιαγραφές που έχουν θέσει φορείς όπως ο ΣΑ και το EFTF θα πρέπει να εντοπιστούν, αλλά αυτές οι δικαιοδοσίες που συμμορφούνται όπως το Τζέρζι θα πρέπει να αναγνωριστούν διεθνώς ως τέτοιες. Αυτό που είναι σημαντικό ότι η κατηγοριοποίηση των δικαιοδοσιών θα πρέπει να εδράζεται επί αντικειμενικών στοιχείων και σχετικής αναλύσεως. Έχοντας αυτό υπόψη μεταξύ άλλων, καλωσορίζουμε τη δυνατότητα να σας δώσουμε πληροφορίες για το Τζέσι. Και το τρόπος θεωρώ ότι η Επιτροπή θα έχει την επιστολή που έστειλε ο Υπουργός Αρμόδιος στις 29 Μαΐου του 2015 και από αποστάλει στον πρόεδρο από τους αρμόδιους υπουργούς Τζένσε και Γκένσε με ημερομηνία 22 Φεβρουαρίου 2016. Η σταματική μας θέση αναφέρεται στις επιστολές και ταιριάζει και με αυτά που περιέγραψε εκπρόσωπο του Γκένζ. Είναι παρόμοια θέση όμω και δεν θα την επαναλάβω. Μια πτυχή που καλύπτεται σε επιστολέ που θα ήθελα να τονίσω εκ νέου είναι η εξή. Η πολιτική καλή γειτονία που επιδιώκεται στι σχέσει μα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Τζέρσι, δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αναγνωρίζει ότι ανήκει στην Ευρώπη. Η επιθυμία να ενισχυθεί αυτή η σχέση περαιτέρω οδήγησε στο να δημιουργηθεί υπηρεσία των χωρών ε, ε, της περιοχής της Μάχης ε, ε, ε, στις και ε, εκπρόσωπο είναι ο κ. Βίλιαμ που είναι εδώ. Και θέλουμε διαθετήσει με τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω σε επίσημο και θεσμικό επίπεδο. Οι υπουργοί επεσκέφθησαν τρει φορέ τι Βρυξέλλε τα δύο χρόνια και τονίζουν στι επιστολέ των Πρόεδρων τη σημασία που προσδίδουμε στην περαιτέρω ε, ανάπτυξη των επαφών με το Ευρωκοινοβούλιο σε αυτό το πλαίσιο διότι και συνομιλίε. Θέλουμε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέματα φορολογικά. Αυτό αναφέρεται στα παρατήματα των επιστολών. Μετά από μια συνάντηση με του υπουργού τον Ιανουάριο, ο Επίτροπο ο κ. Μοσκοβιτσή επένεσε τι νήσου για τη συνεργασία του και θεώρησε ότι σημαντική εταίρη τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω η εθελοντική υποστήριξη τη οδηγία Ευρωπαϊκή Ενώσεω για την φορολόγηση των αποταμιεύσεων και ε, για την φορολόγηση των επιχειρήσεων σύμφωνα με ομάδα δείχνουν ότι θέλουμε συνεργαστούμε. Και η συνεργασία όμω ξεπερνά τα, ξεπερνά τα προλογικά. Θέλουμε να συνεργαστούμε και για την επιβολή κυρώσεων. Αυτό έχει εκτιμηθεί και την Υπηρεσία Εξωτερική Δράσεω. Και αυτό είναι άλλο ένα παράδειγμα επιθυμία συνεργασία. Πριν αναφερθώ στη συμμόρφωση του Τζέσι με τι διάφορε φορολογικέ πρωτοβουλίε που πιστεύω ότι η Επιτροπή τι βρίσκει ενδιαφέρουσε, θα ήθελα να αναφερθώ σε μια πτυχή όσον αφορά το σύστημα φορολογική των επιχειρήσεων. Οι πληροφορίε αναφέρονται στην αλληλογραφία με τον Πρόεδρο που σα προανέφερα. Λοιπόν, το ποσοστό της φορολόγησης είναι 0%, με 10% είναι το ύψιστο ποσοστό για τις εταιρείε που παρέχουν χρηματοστικές υπηρεσίες και τα κέρδη που δίνονται στους μετόχους φορολογούνται στα χέρια των μετόχων στο 20% και είναι το μέγιστο ποσοστό του φόρου εισοδημάτων των ατόμων. Κανένα, ε, δεν υπάρχει κανένα κίνητρο για εξαιρέσει ε, σε άλλους υπουργούς κλπ ε, που να παράγουν ε, σωστή επιβολή των φόρων των εταιρικών. Λοιπόν, είναι απλό το σύστημα των φορολογήσεων και ενίσω δεν χρειάζεται τι αποφάσει φορολογικέ tax rulings που χρειάζονται σε άλλε δικαιοδοσίε. Το 0% φορολογική επιχειρήσεων βασίζεται σε δύο αρχέ. Πρώτα απ' όλα η βασική αρχή τη μη διάκριση μεταξύ των κατοίκων και μη των χωρών που έχουν την έδρα εκεί και δεν έχουν και θεωρείται ότι το σύστημα φορολογήσεων είναι επιβλαβέ. Μετά έχουμε την αρχή τη ουδετερότητα του φόρου που συνδυάζεται με τη διαφάνεια σαν Διεθνές κρηματοστικό Κέντρο το Τζέσι είναι ε, διευκολύνει μάλλον τις επενδύσεις πόρων από όλο τον κόσμο ε, στις ευρωπαϊκές χρηματαγορές και θεωρεί ότι η απόδοση των επενδύσεων πρέπει να φορολογείται στα κράτη που έχουν ε, την έδρα τους οι επενδυτές. Και θα πρέπει λοιπόν να φορολογείται η δραστηριότητα εκεί που λαμβάνει η χώρα. Η κυβέρνηση του Τζέζι να γνωρίζει ότι για να εισπράττεται ο φόρος εκεί που οφείλεται θα πρέπει χώρες οι ενδιαφερόμενε να έχουν τι κατάλληλες πληροφορίε για να κάνουν σωστέ αξιολογήσει. Του με τότε υπόψη το Τζέσι έχει υποστηρίξει πλήρω τη διαφάνεια, την αρχή τη διαφάνεια και είναι στο επίκεντρο στι αποφάσει τη Ευρωπαϊκή Ενώση των ΟΣΑ και των G20. Πιστεύει ότι κάθε δικαιοδοσία μπορεί να καθορίζει τα δικά τη ποσοστά φορολόγηση σύμφωνα με τι δικέ της απαιτήσει, αλλά θα πρέπει να συμμορφώνεται αυτή η δικαιοδοσία και με διεθνεί αρχέ, δίκαιο φορολογικού ανταγωνισμού με διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών. Και αυτό οδηγεί βεβαίω στην περιγραφή τη θέσεω του Τζέσι όσον αφορά αυτό που θεωρούμε ότι είναι βασικό στοιχείο όσον αφορά τη διεθνή καταπολέμηση τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Καταρχά, χρειαζόμαστε ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν ετήσεω. Εμεί ανταλλάσσουμε πληροφορίε κατόπιν αιτήματο σύμφωνα με τι διεθνεί προδιαγραφέ και την πρωτοβουλία του ΟΣΑ του 2002. 38 ανταλλαγές συμφωνίες ανταλλαγή πληροφοριών και διαφόρων άλλων συναφών ε, συμφωνιών έχουν υπογραφεί. 40 εφαρμόζονται συμφωνίες. Από το 2014 το Τζέζι συμμετέχει στην πολυμερή σύμβαση για αμοιβαία διοικητική αρρωγή φορολογικά και μέσω αυτού ανταλλάσσεται πληροφορία με άλλες 22 δικαιοδοσίες. Από το 2009 μέχρι το 2013 το Τζέσι ήταν αντιπρόεδρος της ομάδας ε, του Παγκόσμιου Φόρουμ για τη διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικού σκοπούς και ο φορέας εποπτεύει τη συμμόρφωση με διεθνείς προδιαγραφές. Δεύτερον, η αυτόματη ανταλλαγή των πληροφοριών. Υποστηρίξαμε την πρωτοβολία των G5 για την θέτηση των κοινών προτύπων για την υποβολή εκθέσεων και οθέτησε τι προδιαγραφέ. Υπέγραψε την πολυμερή συμφωνία τη Αρμόδια Αρχή στο Βερολίνο τον Οκτώβριο του 2014. Το Τζέσσι έχει νομοθεσία που εφαρμόζεται και η πρώτη ανταλλαγή των πληροφοριών θα λάβει χώρα το 2017. Το Τζέσσι έχει θέσει αντιπροέδρου του Παγκοσμίου ε, Φόρουμ ομάδων εργασιών ε, και εκεί δείχνει πώς, μπορούμε, πώς συμβάλλουμε μάλλον στην πρωτοβουλία. Μετά τώρα η ιδιοκτησία, η ουσιαστική ιδιοκτησία. Έχουμε μητρό αυτή της ε, ιδιοκτησία, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να εφαρμόσουμε εκεί τη διαφάνεια. Σύμφωνα με την αρμόδια οδηγία, η Παγκόσμια Τράπεζα στην έκθεσή της εντοπίζει ότι το πρότυπο του Τζένσι δημιουργεί τι προποθέσει, ούτω ώστε το μητό των επιχειρήσεων θεωρείται μια βιώσιμη επιλογή για να δίνουμε πληροφορίε για την πραγματική διοκτήση των επιχειρήσεων. Θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση των πληροφοριών του Μητρώου και οι πάροχοι που δίνουν πληροφορίε θα πρέπει επίση να συμμορφούνται με την νομοθεσία και το Μητρό στελεχιώνεται από εκείνου που έχουν την τεχνογνωσία. Το Τζέσι επίση ηγείται στο βαθμό που ε, συμμορφώνεται στη στάση για την καποδολέμηση του ξεπλήματο χρήματο και συμμετέχει στην αρμόδια Task Force. Και παρέχει στην Task Force συστάσει εν γέννη και πρέπει να σημειωθεί ότι το Τζέσι θεωρεί ότι η φοροδιαφυγή ήταν αδίκημα που θεσπίστηκε το 1999 πολλά χρόνια πριν έχει γίνει η σύσταση τη ομάδα κρούση Task Force. Τέταρτον, λοιπόν, τα BEPS ε, συμμορφωνόμαστε και υποστηρίζουμε το πρόγραμμα BEPS και θέλουμε να ενημερωνόμαθα για την πρόοδο για την εφαρμογή των σχετικών δράσεων που απαρτίζουν το πρόγραμμα. Έγκαιρη δράση έγινε για την υποβολή εκθέσεων κατά χώρα σαν φατακέρδια από πολυεθνικές επιχειρήσεις και προς το κάτω ότι θα είναι περιορισμένη η εφαρμογή στους αφορά επιχειρήσεις που εδρεύουν στο Τζέσι. Παρ' όλα αυτά ε, υπάρχει διαβούλευση με, με το χρηματοδοτικό κλάδο για το θέμα αυτό και αναμένεται σπιστή νομοθεσία παρόμοια με αυτή που εφαρμόζει το Ηνωμένο Βασίλειο τελικά μετά τις διαβουλεύσεις. Έχουμε διπλές, ε, λίγες συμφωνίες για τη διπλή φορολόγηση και έτσι δεν έχουμε προβλήματα μετακίνηση των κερδών όπως σας δικαιοδοσίες. Όμως θα εξετάσουμε τι ε, νομοθεσία χρειαζόμαστε για να συμμετάσχουμε στο BEPS όταν θα είναι σαφέστερες οι δράσεις που θα εφαρμοστούν από τους G20 τον ΟΣΑ και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η πρόταση ότι θα πρέπει να φορολογούνται τα κέρδη εκεί που γεννάται η οικονομική δραστηριότητα, που γεννάται το κέρδος, ε, ταιριάζει με την ιστορική μας πολιτική. Θέλουμε τα χρησιμοτικά ιδρύματα όπως οι τράπεζες να έχουν πραγματική φορολογική παρουσία και αυτό αντικατοπτρίζεται στο ότι ο τομέα απασχολεί περίπου 13.000 άτομα και η πρόταση BEPS θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση μα. Πέμπτον, να βοηθήσουμε τι αναπτυσσόμενε χώρε. Το Τζέρσι άμεσα συμμετέχει στι προσπάθειε των αναπτυσσόμενων χωρών μέσω βοηθεία του παρέχει την καταπολέμηση ε, του εγκλήματος. Αυτό αντικατοπτρίζεται στη δίωξη εκείνων που είχαν ανοιχθεί με διαφθορά στην Ιγυρία και στην Κένια πιο πρόσφατα και τον επαναπατρισμό των ε, κλεμμένων ποσών. Σε συζήτηση με κάποιε μη κυβερνητικέ οργανώσει που δραστηριοποιούνται στον τομέα, το Τζέρσι ανέφερε ότι καταρχήν δεν είναι κατά τη αυτόματη ανταλλαγής πληροφοριών και σχετική συμφωνίας επί μία αμοιβαία βάση, ούτε ώστε οι πληροφορίες να παρέχονται στην αναπτυσσόμενη χώρα χωρί αμέσω να πρέπει να εφαρμόσουν αναγκαίε διαδικασίε για να συλλέξουν εκείνε τι πληροφορίε που θα δώσουν ε, ως αντίβαρο. Ελπίζουμε μέσω των εισαγωγικών αυτών σχολείων και των απαντήσεων που θα δώσουμε σε τυχόν ερωτήσει, ότι η Επιτροπή θα αναγνωρίσει και θα αποδεχτεί ότι έχουμε την ίδια αφοσίωση να συμμορφωθούμε με τις σχετικές διεθνεί ε, προδιαγραφές και το πολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και ότι έχουμε πραγματικά συμμορφωθεί με αυτή την δέσμευση που έχουμε αναλάβει. Αυτά και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ καλά, σας ευχαριστώ λοιπόν. Θα δώσω το λόγο στον συγγητή και τους εκπροσώπους των ε, ομάδων. Έχουμε την αρχή ερωταπαντήσεων περίπου πεντάλεπτο η διάρκεια. Συμβουλεύω λοιπόν σε όλους τους παρεμβαίνοντες να είναι όσο πιο λακωνικοί μπορούν στις ερωτήσεις τους και να διευκρινίσουν αν η ερώτηση απευθύνεται στο Τζέρσεϊ, το Γκέρνζε ή και στους ε, δύο και θα ζητούσα από τους εκπροσώπους του Γκέρνζε και του Τζέρσεϊ να φροντίσουν να λαμβάνουν υπόψη τους και το χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους. Εμφανίζεται στο χρονόμετρο. Ναι. Λοιπόν, έχετε το χρονόμετρο που εμφανίζεται ούτως ώστε να τηρούμε το πεντάλεπτο για τις ερωταπαντήσεις καταρχάς τον συνσηγητή τον Γεπ Κόφοντ. Κόφοντ, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Ρομπ Κρέι και τον Κόλιν Πάουελ που ήρθαν εδώ στην Επιτροπή μας σήμερα για να μας εξηγήσουν την κατάσταση στο Γκένσι και στο Τζέρσι. Και που μας εξηγήσατε και πώς συνεργάζεστε μεταξύ σας σχετικά με τα πρότυπα του ΩΣΑ όσον αφορά τα BEPS και την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Η ερώτησή μου θα είναι σύντομη, διότι θα ήθελα να ακούσω τις απαντήσεις σας. Από ό,τι καταλαβαίνω, ένα από τα προβλήματα είναι ότι δεν έχετε πληροφορίες όσον αφορά την επίσημη κυριότητα των επιχειρήσεων που έχουν έδρα στο Γκέρνσι και στο Τζέρσι. Ε, δεν υπάρχουν επιγραμμικά δηλαδή, δεν μπορεί το κοινό να δει τις πληροφορίες αυτές. Ήθελα λοιπόν ε, να βεβαιωθώ ότι ε, οι επενδύσεις των επιχειρήσεων που δεν έχουν έδρα στην... στο Κέρσι και στο Τζέρσι φορολογούνται εκεί όπου κατοικούν οι ιδιοκτήτες των εταιριών. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Και όσον αφορά την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, από ό,τι καταλαβαίνω, και η ερώτηση αυτή απευθύνεται περισσότερο στον Colin Powell, είσαστε διατεθειμένοι να ε, προσορίσετε στο καθεστώς αυτό, της αυτόματης ανταλλαγής. Και θα ήθελα να μου εξηγήσετε ποιες είναι οι επιφυλάξεις αυτό το θέμα αυτό. Και τέλος, ίσως να μην καταλαβαίνω το καθεστώς εταιρικής φορολογικής σας ε, έχετε συντελεστεί 0% και παρόλα αυτά υποστηρίζετε ότι είσαστε υπέρ του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και της καταπολέμησης της φοροαποφυγής. Πώς συμμορφώνεται ο μηδενικός συντελεστής με την καταπολέμηση της φοροαποφυγής. Ε, θα με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω ποιος θέλει να απαντήσει. Και οι δύο. Ο κύριος Πάουελ. Ευχαριστώ πολύ, ε, Πρόεδρε, και σε ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Επιτρέψτε μου να αρχίσω με το θέμα της ιδιοκτησίας εταιριών. Πώς έχει η κατάσταση στο Τζέρζι και είναι ενδεικτικό. Έχουμε ένα μητρό επιχειρήσεων που έχει προνομιούχες προφορίες για το ιδιοκτησιακό καθεστώς που διαφέρει αυτό σημαντικά από άλλες δικαιοδοσίες. Έχουμε λοιπόν αυτό το μητρό που επικοινώνεται σε μεγάλο βαθμό από εκείνους που παίρνουν τις προφορίες. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι ότι δεχόμαστε ό,τι προφόρηση μας δίνουν εταιρείε, το ψάχνουμε οι, οι άλλοι οργανισμοί. Και επίση mm. Υποστηρίζουμε αυτή τη διαδικασία για να βεβαιωθούμε ότι οι προφορίες αυτές είναι σωστές, ακριβείς και επίκαιρες και σε τακτά χρονικά διαστήματα τα αναθεωρούμε και εκείνοι που διαχειρίζονται τι εταιρείε έχουν και εποπτεία, έχουν και κανόνες και ε, ξέρουμε ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης. Και αν δεν γίνεται αυτή ε, η ε, δουλειά αποτελεσματικά υπάρχει κίνδυνος να διωχθούν και να χάσουν και την άδεια της ε, επιχείρησης και να την κλείσουν. Δηλαδή το μητρό αυτό έχει στοιχεία πάρα πολύ ακριβή, ε, πάρα πολύ επίκαιρα και πάρα πολύ σωστά. Ε, το μόνο πρόβλημα που έχουμε διαπιστώσει μέχρι σήμερα είναι το εξής. Πρώτη μας προτεραιότητα είναι οι πληροφορίες να διατίθενται ε, στις φορολογικές και στις ε, αρχές επιβολής του νόμου. Ε, σωστές, ακριβείς πληροφορίες και επίκαιρες. Ενημερωμένα στοιχεία δηλαδή. Αυτό το κάνουμε με τρόπο πάρα πολύ αποτελεσματικό. Εάν η επέκταση της διαδικασίας αυτής τελικά θα πρέπει να είναι η δημοσίευση για το κοινό, κοιτάμε τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές, τι πρέπει να γίνει. Ε, με την οδηγία, ε, την ε, τέταρτη οδηγία τη σχετική δεν απαιτεί δημοσιοποίηση στο ευρύ κοινό και υπάρχουν διάφορες συστάσεις διεθνείς που δεν προβλέπουν. Δεν επιμένουν καν να υπάρχει ένα κεντρικό μητρό. Πάντως, εμείς ακολουθούμε αυτές τις προδιαγραφές και όπως εξελίσσονται τις υιοθετούμε και να είστε βέβαιοι ότι και το Τζέρσι θα δώσει συνέχεια σε όλα αυτά που λέτε. Το Γκένσι. Θα ήθελα να προσθέσω λίγο ε, τη σκοπιά τη δική μας ε, για το θέμα της πραγματικής ιδιοκτησίας μιας επιχείρησης. Το Γκένσι δεν έχει κεντρικό μητρό επιχειρήσεων. Η κατάσταση λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με την ε, δυνατότητα πρόσβαση στα στοιχεία είναι πολύ αντίστοιχη με το Τζέρσι. Προηγουμένω σα μίλησα για την νομοθεσία ε, που ε, ανάγεται στο 2000 που έχει να κάνει ε, με τα καταπιστεύματα που θα πρέπει να γνωρίζουν ποιοι είναι οι πελάτες τους σύμφωνα με την δέουσα επιμέλεια για την καταπολέμηση της νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε, το ξέπλυμα δηλαδή χρήματο. Υπάρχουν παρόμοιε διατάξει με το Τζέρσεϊ, δηλαδή αν θέλουμε εμεί να έχουμε πρόσβαση σε προνομιούχα στοιχεία που το έχουμε κάνει ε, ε, μετά από ε, ανταλλαγή πληροφοριών και συμφωνίες που είχαμε σχετικές με φορολογικές αρχές και μας ζήτησαν τα στοιχεία αυτά τα δώσαμε γιατί μπορούμε να τα διαβιβάζουμε. Σε ό,τι αφορά τη βασική ερώτηση που έχει να κάνει με το κεντρικό ε, μητρό έχουμε τον ίδιο στόχο με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θα πρέπει σε πραγματικό χρόνο να έχουμε πρόσβαση σε ακριβή στοιχεία. Ε, βέβαια ένα μητρό αυτό θα το διευκόλυνε. Κάνουμε τέτοια βήματα ε, για να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή, τα είπα και προηγουμένως και στον Γκένζεϊ θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα ασφαλές, ε, ενοποιημένο, τοπικό, με ένα ε, συγκεκριμένο πιστοποιημένο και διαπιστευμένο σύνδεσμο που θα ε, παρέχει πρόσβαση. Είμαστε καθοδόν και το 2017 αναμένεται να γίνουν συστάσεις στη Βουλή μας για να υποβληθούν προς έγκριση. Αυτά. Ναι, ευχαριστώ. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, λέει ο Πρόεδρο. Θα επανέλθουμε και με άλλε ερωτήσει, ιδιαίτερα αυτό το πρόβλημα ε, του μηδενικού φορολογικού συντελεστή. Ε, ε είμαι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν και άλλε ερωτήσει σχετικά. Ας προσπαθήσουμε να τηρούμε το πεντάλεπτο για την ερώτηση και την απάντηση, παρακαλώ. Σύντομε ερωτήσει και σύντομε απαντήσει. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Τώρα, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, η κυρία Ντανούτα Χιούμπνερ. Σύντομη, παρακαλώ να είστε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Στην επάντηση της επιστολής που απέστειλε σε εσά ο κ. Λαμασούρ, είπατε ότι η Διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ενώσης για Διοικητική Συνεργασία και Ανταλλαγή Πληροφοριών δεν ισχύει στη δική σας νομοθεσία. Πρόσφατα ακούσαμε ότι κάποιες μικρές χώρες όπως Ανδόρα, το Λίχτενστάιν και το Μονακό πιθανότητα στο μέλλον έχουν υπογράψει ε, συμβάσεις για ανταλλαγή πληροφοριών με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Το εξετάσατε αυτό το ενδεχόμενο. Θέλω να ξέρω περισσότερο για τα νομικά μέσα που διαθέτει στην νομοθεσία για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερη ερώτηση έχουμε συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του πακέτου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Αντιμπέψ. Δεν στοχεύουμε στην αντιγραφή των BEPS, αλλά θέλουμε να καλύψουμε και την ανάγκη που τονίζεται εδώ να έχουμε καλή ισορροπία μεταξύ καλύψεως των αναγκών της ενιαίας αγοράς και της συμμόρφωσής μας με διεθνείς προδιαγραφές και μάλιστα να τον εσείς πώς το βλέπετε. Και σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της ενιαίας αγοράς. Και σε σχέση με τη θέση που έχετε για τα διάφορα εργαλεία αντιπέψ. Δεν ξέρω ποια είναι θέση σας. Ο κ. Γκρέι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για το πρώτο ερώτημα. Το Γκένζι επί σειρά ετών από το 2005 έχει εφαρμόσει συμφωνίες με κράτη μέσα Ευρωπαϊκής Ενώσης που αντιστοιχούν στην οδηγία για τις αποταμιεύσεις. Και που στο τέλος του περασμένου έτους αποστήλαμε επιστολές σε όλα τα κράτη-μέλη αναφέροντας την πρόθεσή μας να σταματήσει η εφαρμογή της ε, οδηγίας και να μπούμε στις προδιαγραφές για την υποβολή εκθέσεων. Από την αρχή του επομένου έτους θα ανταλλάσσουμε πληροφορίες που αφορούν το 2016. Για αρκετά χρόνια λοιπόν είχαμε αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και αυτό σύμφωνα με τις συμφωνίες που αντιστοιχούν στην οδηγία για τις αποταμιεύσεις. Και από του χρόνου θα ανταλλάσσουμε πληροφορίες με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως επί της βάσης των προδιαγραφών για υποβολή πληροφοριών, των κοινών προδιαγραφών για ανταλλαγή πληροφοριών. Πιστεύω ότι έτσι απάντησα. Ο κύριος ε, Πάουλ τι έχει να πει. Απλώς να συνεχίσω κι εγώ το δεύτερο ερώτημα το αντι Είπαμε ότι θέλουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα BEPS και το Jersey και το Genzy αλλά όπως προανέφερα, επί σειρά ετών ακολουθήσαμε μια πολιτική καλής γειτονίας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σεβόμεθα τα όσα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όσον αφορά τα προγράμματα BEPS-ANTI-BEPS, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Θα εξετάσουμε τις λεπτομέρειες. Εν γέννη όμως, η γενική μας άποψη είναι η εξής. Χρειάζεται διεθνή συμμόρφωση. Πολύ σημαντική αρχή αυτή η διεθνής συνέπεια. Όχι μόνο για τις επιχειρήσεις και τα χρηματοστατικά ιδρύματα και για τις κυβερνήσεις. Εφαρμόζουμε τα BEPS, θέλουμε να εφαρμόσουμε πολιτική καλής γειτονίας, ταυτοχρόνως επιδιώκουμε συμμόρφωση, συνέπεια και σαφή γενική εικόνα για την όλη κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Η Άννα Γκόμες έχει το λόγο. Μπορείτε παρακαλώ να μου εξηγήσετε τι είδους δικαιοσύνη υπάρχει σε ένα σύστημα που φορολογεί ε, άτομα, δεν φορολογεί όμως τις επιχειρήσεις. Και εάν κάθε κυβέρνηση το έκανε αυτό, πού θα βρισκόμασταν όσον αφορά τις ανισότητες στον κόσμο. Είπατε ότι εδώ και αρκετά χρόνια δεν ε, έχετε φορολογικές αποφάσεις τύπου tax rulings αλλά προβλέπονται παρεκκλήσεις ε, ή ειδικά ωφέλη σε άτομα, σε, στα άτομα που φορολογούνται με 20%. Και με τι κριτήρια γίνεται αυτό και υπάρχει κάποιος έλεγχος, γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν έχετε κοινοβούλια δικά σας, έτσι δεν είναι. Προβλέπονται λοιπόν τέτοιε ε, παρεκκλήσει ε, ή ειδική μεταχείριση ατόμων όπω συμβαίνει αλλού. Και όσον αφορά την πραγματική κυριότητα των εταιριών, κατάλαβα από τον κύριο Γκρέι ότι ζητά, ζητάτε να συγκεντρώνονται οι σχετικέ πληροφορίε. Αυτέ όμω πού συγκεντρώνονται οι εταιρείε, φροντίζουν γι' αυτό ή υπάρχει κάποιο κεντρικό μητρό. Και οι αρχέ επιβολή του νόμου έχουν πρόσβαση στι πληροφορίε αυτέ. και μπορεί και το κοινό να έχει πρόσβαση στα μητρώα αυτά σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο θεμητό συμφέρον και όσον αφορά τα ιδρύματα και τα καταπιστεύματα. Υπάρχει υποχρεωτική καταχώρηση των πραγματικών ιδιοκτητών. και τι διαφορά υπάρχει ανάμεσα σε, σε εσά, σε τον Γκέντσι και τον Τζέρσι και το ε, Γιβραλτάρι ή ε, τις Βερμούδες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλές ερωτήσεις ακούστηκαν. Δεν ξέρω αν μπορώ να περιοριστώ σε πέντε λεπτά. Ας ξεκινήσω από την πρώτη ερώτηση. Σχετικά με το ότι φορολογούμε ε, τα άτομα, όχι όμως τις επιχειρήσεις. Φορολογούμε πολλές επιχειρήσεις, διότι Παρότι έχουμε μηδενικό συντελεστή φορολογία, ε, εφαρμόζεται το 10% σε εταιρείε ε, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Και καθότι είμαστε Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Κέντρο, καταλαβαίνετε ότι αυτός ο τομέας είναι πολύ σημαντικός όσον αφορά τη συνεισφορά στα φορολογικά μας έσοδα. Μάλιστα, από τα συνολικά ε, φορολογικά έσοδα, η αναλογία των φόρων από εταιρείε ε, αντιστοιχεί σε αυτό σε άλλες χώρες, ε, γύρω στο 25%. Δηλαδή βρισκόμαστε περίπου στο ίδιο επίπεδο με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο μηδενικός φορολογικός συντελεστής ισχύει σε επιχειρήσεις που ανήκουν σε κατοίκους των ε, νησιών μας. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, ε, φορολογούνται οι επιχειρήσεις ε, με τους κανόνες αυτούς. Και να δώσω το λόγο στον συνάδελφο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσω στη δεύτερη ερώτηση που είχε να κάνει με το πώς φορολογούμε τα άτομα. Όσον αφορά τον Γκένση, και νομίζω ότι και το Τζέρσι εφαρμόζει παρόμοιο σύστημα, το 1920 είχαμε τους πρώτες ε, κανόνες που βασίστηκαν σε μεγάλο βαθμό στο ισχύον βρετανικό σύστημα. Όσον αφορά λοιπόν τη φορολογία ατόμων, δεν έχει αλλάξει δραματικά έκτοτε. Έχουμε σύστημα κατοίκων, δηλαδή ε, τα άτομα φορολογούνται ανάλογα με το αν είναι κάτοικοι ή όχι του νησιού και στο ένα άκρο έχουμε έναν μη κάτοικο που φορολογείται ε, για κάποια εισοδήματα όπως ε, είναι ε, η απασχόληση ή τα ενίκια ακινήτων στο νησί. Από την άλλη έχουμε κατοίκους του νησιού μας που φορολογούνται για τα έσοδά τους σε όλο τον κόσμο προβλέπουμε κάποιες δυνατότητες ε, για άτομα όσον αφορά τους ε, τόκους κλπ. Και έχουμε επίσης ε, και ένα σύστημα οροφής, διότι το, η τοπική μας κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι όταν κάποιο άτομο έχει συνεισφέρει αρκετά στα φορολογικά έσοδα του νησιού, υπάρχει ανώτατο όριο. Δηλαδή κάποια άτομα δεν μπορούν να πληρώσουν πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσό σε φόρους ε, και αυτό ισχύει σε όλους και νομίζω ότι ε, σε 30 ή 40 άτομα εφαρμόζεται τελικά αυτό το ανώτατο όριο. Αυτό όσον αφορά τον προσωπικό φόρο. Και όσον αφορά το Μητρό ε, Ιδρυμάτων, ναι, η τελευταία ερώτηση έχει να κάνει με τις εταιρείες καταπιστευματικής διαχείρισης. Όπως και οι περισσότερες άλλες δικαιοδοσίες, δεν έχουμε κεντρικό μητρό, αλλά η διαφορά μας από άλλες δικαιοδοσίες είναι, όπως είπα νωρίτερα, ότι έχουμε πολύ αυστηρό καθεστώς για την αδειοδότηση των ε, επιχειρήσεων ε, καταπιστευματικής διαχείρισης ε, και ε, παροχής σχετικών υπηρεσιών. Όποτε λοιπόν έχουμε λάβει αίτημα για πληροφορίες από τις χώρες με τις οποίες έχουμε συμφωνίες ανταλλαγής πληροφοριών, μπορέσαμε πολύ γρήγορα να τους δώσουμε στοιχεία για την πραγματική κυριότητα ε, και τα πρόσωπα που συμμετέχουν ε, σε αυτές τις εταιρείες ε, καταπιστευτικής διαχείρισης. Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά από τις περισσότερες, αν όχι όλες τις άλλες δικαιοδοσίες. Εάν υπάρξει διεθνές πρότυπο, και φυσικά έχουμε κοιτάξει τις απαιτήσει της οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομων εξόδων, και επειδή θέλουμε να έχουμε ε, καλές ε, σχέσεις γειτονιές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σίγουρα θα ανταποκριθούμε. Ε, Βρίσκαστε μπροστά από πολλούς άλλους και του γειτονά σας. Στο θέμα αυτό είμαστε σαν δίδυμοι. Καλώς, ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο Ασλή Φόξ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κρέι και τον κύριο Πάουερ που ήρθαν σήμερα στην συνεδρίασή μας. Ξεκαθαρίσατε στην επιστολή σας όταν δεχθήκατε να έρθετε εδώ ότι τα νησιά της Μάχης ήταν πάρα πολύ δραστήρια στις διεθνείς ε, καινοτομίες και πρωτοβουλίες κατά της ε, φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Νωρίς μάλιστα ε, υιοθέτησαν τα νησιά αυτά ε, τις διεθνεί προδιαγραφέ για ανταλλαγή Πληροφοριών. Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω και του δύο. Ε, λέγουν ότι οι δικαιοδοσίες τους ε, συμμορφώνται προς τη χρηστή διακυβέρνηση και σε Ευρωπαϊκέ και διεθνεί προδιαγραφέ. Θέλω να του ζητήσω τη συμβουλή του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί, μπορεί να βοηθηθεί να δει και να καταλάβει περισσότερο τη διαφορά ανάμεσα στις δικαιοδοσίες που συμμορφώνονται και εκείνες που αρνούνται να το πράξουν. Πώς μπορούμε να τη βοηθήσουμε να φωτιστεί. Ευχαριστώ ε, για την ερώτηση αυτή. Είναι σημαντικό το ζήτημα. Καλώς ορίσαμε την περιγραφή του Γκέρνζε και του Τζέρζε που έκανε ο κύριος Μοσκοβισή, ο Επίτροπος, ότι είναι δικαιοδοσίες που ε, συνεργάζονται και ως εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εμείς έτσι το βλέπουμε. Έχουμε μια εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα μας βοηθούσε αν αυτή η αναγνώριση ήταν πιο συνεπής και πιο συνεχής. Υποστηρίζουμε την προσέγγιση της ε, του 2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις συστάσεις για το πώς ορίζεται η χρηστή διακυβέρνηση από τρίτες χώρες σε σχέση με ε, την ε, προσήλωση σε διεθνείς προδιαγραφές και τις ίδιες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα όπως ορίζονται από τον κώδικα διοντολογίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό υποστηρίζουμε και την προσέγγιση στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 28 Ιανουαρίου ενεστώτος έτους για τα διαφανή κριτήρια και τις ε, διεθνείς ε, και ευρωπαϊκές συμφωνίες. Αυτή η διάκριση αυτό τον καιρό είναι ε, κάτι που παρεμποδίζεται γιατί η συνεργασία μας μπορεί να σκιαστεί από τη συζήτηση που γίνεται για τους φορολογικούς συντελεστές. Συνεχίζονται οι συζητήσεις και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο για μια ελάχιστη αποτελεσματική φορολόγηση. Αλλά αυτή τη στιγμή μεταξύ κρατών μελών δεν επικρατεί συνένεση για το συγκεκριμένο θέμα ακόμα, ούτε καν για την εσωτερική πολιτική. Οι φορολογικοί συντελεστέ δεν είναι από τα κριτήρια που συνιστά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωση του Ιανουαρίου. Ξέρουμε και μια ε, έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε το Δεκέμβριο, ούτε και αναφέρονται οι φορολογικοί συντελεστές. Τα κράτη-μέλη έχουν κάποια κριτήρια ε, ε, ε, λέγεται CFC αυτή η νομοθεσία για τις ελεγχόμενες ε, ξένες επιχειρήσεις. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με τους φορολογικούς συντελεστές αλλά δεν θα πρέπει αυτές οι δικαιοδοσίες να εγγράφονται σε μαύρες λίστες γιατί αυτό είναι εκτός της σημερινής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, εκπρόσωπος του Ναι, στο τελευταίο αυτό που είπε ο συνάδελφος θα είχα να προσθέσω το εξής προσεγγίσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκείνες τις δικαιοδοσίες που ακόμα ε, μας έχουν σε μαύρη λίστα uh, για να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε και στον διαδραστικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να γίνεται πιο σαφής διάκριση ανάμεσα σε εκείνες ε, τις χώρες που έχουν μαύρες λίστες για τα σύψη ή ε, για τις χώρες που δεν συνεργάζονται. Ελπίζω τα κράτη-μέλη γενικά να ακολουθήσουν την προσέγγιση που έχει ακολουθήσει η Ιταλία στις αρχές του έτους, που έχει βγάλει από τη μαύρη λίστα ε, για τους φορολογικούς συντελεστές νησιά και λέει ότι αυτή η νομοθεσία αφορά οποιαδήποτε χώρα που δεν ε, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις. Πολλές δικαιοδοσίες και μεταξύ αυτών πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν νομοθεσία για τη φορολόγηση των ξένων εταιριών, αλλά δεν δημοσιεύουν μαύρες λίστες ε, με άλλες δικαιοδοσίες που δεν το εφαρμόζουν, γιατί δίνουν την εντύπωση ότι αν έχεις μια τέτοια μαύρη λίστα, οι χώρες αυτές αθετούν τις υποχρεώσεις τους, ε, ε, τις ευθύνες τους και δεν σέβονται τη συνεργασία. Και ελπίζουμε τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναγνωρίσουν περισσότερο δημοσίως ε, τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων που έχουν γίνει από διεθνείς οργανισμούς όπως είναι το Παγκόσμιο Φόρουμ Διαφάνειας ε, και άλλες εταιρείες και άλλα funds ε, που κατατάσσουν και την Γκέρζε και την Τζέρζε σε υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης με τις διεθνείς προδιαγραφές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Κόρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τους δύο κυρίους που ήρθαν στην Επιτροπή μας. Αναφερθήκατε και δύο στη διαφάνεια, επανειλημμένα, και στην φορολογική ουδετερότητα. Και έχω σχετικά κάποιες ερωτήσεις για τη διαφάνεια πρώτα απ' όλα. Φαίνεστε ενθουσιώδης όσον αφορά τις διεθνείς ε, συστάσεις. Για τη δημόσια υποβολή εκθέσεων κατά χώρα, πέρα από τα όσα προτείνει ο ΣΑ, ποια είναι η υπόψή σας Είσαστε ακόμα ενθουσιώδεις για μια τέτοια, τέτοιου είδους διαφάνεια. Από ό,τι κατάλαβα, το Τζέσι και το Γκένσι δεν έχουν δεν καλύπτουν την, το απόρριτο των τραπεζών με βάση το ποινικό δίκαιο. Όμως το απόρριτο καλύπτεται μέσω ιδρυμάτων, καταπιστευμάτων κλπ. Μπορείτε να μας πείτε σχετικά με αυτά ποια θα είναι η πολιτική σας. Μάλιστα όταν λέτε ότι θέλετε να συμμορφωθείτε και στις προσπάθει... με τις προσπάθειες που καταβάλουμε εμείς για τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή. Η δικαιοδοσία των ίσων χρησιμοποιείται από τι επιχειρήσει του Ηνωμένου Βασιλείου, ώστε να εντοπίζουν εκεί τι χρηματοστικέ δραστηριότητε. Και υπάρχουν κανόνε του Ηνωμένου Βασιλείου για ελεγχόμενε ξένες επιχειρήσει. Οι εταιρείε που είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να δημιουργήσουν ε, χρηματοδοτικέ εταιρείε στο Γκένσε και στο Τζέσε και να δανείζουν σε ξένες εταιρείες και πληρώνουν μόνο όσον αφορά τους φόρο. 5% ή 0% καμιά φορά βάσει της δικής σας νομοθεσίας. Μου ανταξηγήσετε. Αυτό πώς συνδυάζεται με την έκκλησή σας ε, περί φορολογικής ουδετερότητας. Ευχαριστώ κόρα, Mr. ο κύριος Πάουλ μάλλον. Θα ήθελα να αναφερθώ στη διαφάνεια. Σε αυτά που είπαμε, δείξαμε ότι θέλουμε να εφαρμόσουμε τα προγράμματα BEPS. Και συμμετείχαμε και στην υποβολή εκθέσεων κατά τα χώρα. Έχουμε δρομολογήσει σχετική νομοθεσία. Θα εφαρμοστεί τάχιστα. για την αποκάλυψη στοιχείων και το απόρριτο των στοιχείων και τη δημοσιοποίησή τους. Το εξετάζουμε το θέμα. Θέλουμε να δούμε ποιο διεθνές πρότυπο θα επικρατήσει και τι θα γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό περιμένουμε με ενδιαφέρον αυτό που θα προκύψει σύντομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί από τα κράτη-μέλη. Η θέση μας είναι θέση σεβασμού και συμμόρφωσης με τη διεθνή θέση. Να διορθώσω κάτι που αναφέρθηκε για τα στοιχεία, για το απόρριτο τραπεζόν, τραπεζών. Το Τζέσι και το Γκένσι δεν έχουν νομοθεσία για το απόρριτο τραπεζών, όπως υπάρχει σε πολλές άλλες χώρες για το τραπεζικό απόρριτο. Έχουμε διευθετήσεις περιπιστευτικότητας όσον αφορά τα τραπεζικά στοιχεία, όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο και στα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είναι εμπιστευτικότητα που σχετίζεται με την προστασία του ατόμου, των προσωπικών πληροφοριών. Η κυρία που έβαλε την ερώτηση διετείνεται ότι ε, είναι απόλυτα τα στοιχεία που αφορούν τα καταπιστεύματα. Ε, δεν ισχύει μεγαλύτερη μυστικότητα για αυτά από ό,τι έτσι επιχειρήσεις. Με τη σωστή νομοθεσία και τη σωστή πολιτική όπως έχουμε είναι διαφανής η κατάσταση για τα καταπιστεύματα όπως και τις επιχειρήσεις. Αναγνωρίζουμε όμως ότι υπάρχει κάποια δυσκολία. Συνήθως με το αστικό δίκαιο όσον αφορά τα καταπιστεύματα και τι καλύπτει αυτή η έννοια. Στην νομοθεσία μας τι κάναμε. Έχουμε κάνει διαβήματα σε διάφορες νομοθεσίες, κάναμε και παρουσιάσεις. Πήγαμε στο Ελσίνκι, στη Στοκχόλμη, στην Κοπενχάγη, πήγαμε στη Ρίγα για να κάνουμε παρουσιάσεις. Θέλουμε να κάνουμε παρουσιάσεις και στο Παρίσι και στα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, αν το επιθυμούν. Θέλουμε να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια ακριβώς ποια είναι η έννοια του καταπιστεύματος για μας και δεν είναι κάτι τόσο ε, αδιαφανές όπως πιστεύουν κάποιοι. Κυρίως εκείνοι που δεν κατανοούν πλήρω την έννοια, πλήρως την έννοια αυτή. Λοιπόν, αν έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε αυτή τη διευκρίνηση είναι ευπρόσδεκτη για τις ε, βρετανικές επιχειρήσεις. Θα προσπαθήσω λοιπόν να συμμορφωθώ με τα χρονικά μου όρια, να καλύψω τα αναπομένοντα στοιχεία, αθρηστικά, διότι αφορούν το ίδιο ζήτημα. Δηλαδή ανταλλαγή πληροφοριών με χώρες που έχουν θεμητή ανάγκη για τις πληροφορίες. Τις χρειάζονται ούτω ώστε να εφαρμόσει σωστά η νομοθεσία τους για τη φορολογία. Αυτό ισχύει και για το Ηνωμένο Βασίλειο και για άλλες νομοθεσίες που ζητούν πληροφορίες για κάποια εταιρεία στο Γκέντζε ή καταπίστευμα που δραστηριοποιείται στο Γκένζε. Θα χρησιμοποιήσω το Ηνωμένο Βασίλειο σαν παράδειγμα. Έχουμε συμφωνία διπλής φορολόγησης με το Ηνωμένο Βασίλειο από τη δεκαετία του 50. Συμπεριλαμβάνει και ανταλλαγή πληροφοριών στη σχετική διάταξη. Έχουμε συμφωνία για ανταλλαγή πληροφοριών τα φορολογικά με το Ηνωμένο Βασίλειο. Και έχουμε και διακυβερνητική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο που συνήφθη πρόσφατα για ε, τις πληροφορίες και θα μπούμε και στα, στα πρότυπα για την ε, ανταλλαγή πληροφοριών ε, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο από του χρόνου. Έχουμε διάφορα, διάφορους μηχανισμούς. Αν το Ηνωμένο Βασίλειο ή κάποια άλλη χώρα χρειάζεται πληροφορίες, ούτω ώστε να καλύψει ανάγκες που έχει για την καταπολέμηση φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής κλπ από κάποιον από τους κατοίκους τους, τότε μπορούν οι χώρες να πάρουν τις πληροφορίες από τον Γκένζε. Και το Παγκόσμιο Φόρουμ, το ΩΣΑ, επιστώσει ότι το Γκένζι συμμορφώνεται όταν δέχεται τη αιτήματα. συμπληρώσω την ερώτησή σα. Στην αρχή, στην παρέμβασή σα, ένα από του δυο σα, είπατε κάτι. Είπατε ότι έχετε διμερείς φορολογικές συμβάσεις με 23 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Το περιεχόμενο των συμφωνιών είναι το ίδιο όπως στη συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο ή είναι κάτι διαφορετικό. Απάντηση. Ναι, οι συμφωνίες που ανέφερα είναι για πληροφορίες για τα φορολογικά. Έχουμε 60 συμφωνίες με χώρες του κόσμου και 23 από αυτές Τη συμφωνίες αφορούν κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ενώση συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπάρχουν μικροδιαφορές στη διατύπωση, αλλά ουσιαστικά είναι η ίδια συμφωνία. Ευχαριστώ. Η Παλώμα Λόπεθ από την Ενωτική Αριστερά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μιλήσω ισπανικά. Πρώτον, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και τη συμμετοχή σας σήμερα στην Επιτροπή μας. Η σημερινή και αυριανή συνάντηση μας επιτρέπουν να δούμε μια ενδιαφέρουσα σκοπιά. Δηλαδή, πώς η φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή ε, δεν αφορά αφηρημένα μεγάλες πολυεθνικές, αλλά έχει ονοματεπώνυμο εκείνων που σχεδιάζουν μια προσωπική φορολογική στρατηγική μαζί με κάποιες εταιρείες που ελέγχουν με τη βοήθεια των μεγάλων ε, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Τελικά, οι φορολογικές συμφωνίες των μεγάλων πολυεθνικών δεν είναι παρά μόνο ένας κρίκος σε μια συνολική αλυσίδα που χρηματοδοτεί την αναδιανομή του εισοδήματος ε, που παράγουν οι εργαζόμενοι στους μεγάλους ραντιέριδες και σε offshore ε, όπως τα δικά σας νησιά πρωταγωνιστούν. Με εκπλήσει το γεγονός ότι απορρίψατε επανειλημμένα στις δικαιοδοσίες σας να ε, θεωρούνται φορολογική παράδειση. Μα πώς αλλιώς να τα αποκαλέσουμε αυτά τα εδάφη όπου η πλειονότητα των επιχειρήσεων πληρώνουν φόρο μηδενικό επιχειρήσεων και ούτε ε, τα μερίσματα φορολογούνται σε διεθνείς δικαιούχους είτε σε εταιρείε. Περί αυτού πρόκειται ακριβώς. Δηλαδή δεν πληρώνουν φόρο οι άνθρωποι και ούτε υπάρχει δημόσιο μητρό που να είναι προσβάσιμο σε τρίτους. Ε, είτε είναι φυσικά πρόσωπα είτε νομικά πρόσωπα για την ιδιοκτησία των επιχειρήσεων, για τα κέρδη και τους ισολογισμούς. Και οι εταιρείε ε, και οι αρχές τι έκαναν για να απαντήσουν στη χρηματοπιστωτική κρίση. Έφτιαξαν νέα σκοτεινά ε, κατασκευάσματα όπως είναι τα καταπιστεύματα, τα ιδρύματα για να καλύπτουν ε, κάποιες πομπές των κρατών του Περσικού κόλπου και της Κίνας. Ε, τα έχετε κάνει πλακάκια με την χρηματοπιστωτική ε, βιομηχανία στη Βρετανία και χρειάζονται επιπλέον εξηγήσει από αυτέ που είστε ε, διατεθειμένοι να δώσετε και από τη δικαιοσύνη. Αυτό είναι θετικό, αλλά θέλουμε συγκεκριμένε δράσει που να αποδεικνύουν την επιθυμία συνεργασία και όχι μια αυτόματη απάντηση στα σκάνδαλα φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή που ζήσαμε στο παρελθόν. Ειλικρινά, ο διάλογο φτάνει πια. Πάρα πολλά χρόνια συζητάμε, συζητάμε και παρόλα αυτά λίγες είναι οι ελλαγές που έχουν γίνει. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Θεωρείτε ότι τα ενεργητικά ε, των νήσων που είναι ε, χιλιάδες, εκατομμύρια ευρώ έχουν καμία σχέση με οικονομική δραστηριότητα μιας περιφέρειας που έχει ε, εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους. Έχετε στοιχεία, ε, ποσοστά, πόσο είναι οι ξένοι που έχουν στοιχεία ενεργητικού στο Τζένστη και θα μπορούσατε να μας τα αναλύσετε ανά χώρα και ανά ε, ποσό. Ποιο ποσοστό χρηματοπιστωτικής συναλλαγής γίνεται ενδομιλικά ή σε εταιρείε που έχουν τους ίδιους ιδιοκτήτες. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ότι όταν είναι τόσο κοντά το City του Λονδίνου που είναι σημαντικό χρηματοπιστωτικό κέντρο και οι μεγάλες πολυεθνικές να υπάρχει ένα τέτοιο ε, χρηματοπιστωτικό κέντρο τόσο μεγάλο εάν δεν υπάρχει συνενοχή και ε, συγκάλυψη από τις Βρετανικές αρχές. Και τι γίνεται με τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Συνεργάζονται, θα εγκρίνουν ε, τον αντίστοιχο κανονισμό για τη φορολογία των επιχειρήσεων. Αλλιώς θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να δικαιολογήσουμε πώς δεν θα βάλουμε κυρώσεις ή βέτο ε, στις διάφορες ε, κομπίνες που γίνονται εκεί στα νησιά σας μέχρι να, μην, να διευκρινιστεί αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Τι ερώτηση ήταν αυτή τόσο ε, μακροσκελής, μήπως μπορείτε να απαντήσετε πιο σύντομα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Όπως σας είπα στα εισαγωγικά μου σχόλια, το Γκέρντζε θελοντικά συνεργάζεται με το, την ομάδα για τον κώδικα δεοντολογίας και ε, δώσαμε το σύστημά μας στο φορολογικό να εξεταστεί, να ελεγχτεί και βρέθηκαν πολλά στοιχεία επιζήμια τα οποία εμείς ε, όλα τα αναθεωρήσαμε και τα καταργήσαμε χωρίς καμία εξαίρεση. Και τώρα υπάρχει ένα ε, σύστημα 0, 10 και 20% φορολογικός ε, συντελεστής και πάλι αναθεωρείται το σύστημά μας ε, και ο μηδενικός φορολογικός συντελεστής από μόνος του δεν θεωρείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το, την ομάδα του κώδικα διοντολογίας ως επιβλαβής. Το θέμα που ρώτησε η κυρία έχει να κάνει με την κατάχρηση των φορολογικών καθεστώτων αλλού, απανταχού της γης. Ε, αλλά το θέμα που το λύνει αυτό είναι η παροχή πληροφοριών και κινδυνεύω λίγο να ε, ακούγομαι σαν να έχει κολλήσει η βελόνα, αλλά το Γκένζι έχει πολύ καλές επιδόσεις στη συνεργασία με τις διεθνείς προδιαγραφές σε σχέση με τη διαφάνεια και την ανταλλαγή προφοριών, διότι σε τελική ανάλυση ο μόνος τρόπος μια χώρα να μπορέσει να επιβάλλει την ίδια της στην νομοθεσία και να φορολογήσει εκείνους που φοροδιαφεύγουν, που θα έπρεπε να φορολογούνται στην επικράτεια, είναι να έχει την προφορία για να μπορεί να το πράττει. Οι περισσότεροι φορολογούμενοι στα περισσότερα κράτη ε, είναι ε, νομοταγής. Ε, περί τίνος πρόκειται εδώ. Ελπίζουμε ένα μικρό κλάσμα πληθυσμού και κρατών που επιλέγουν για τους δικούς του λόγους να παρανομούν και να φοροδιαφεύγουν, να φοροαποφεύγουν ή με επιθετικό τρόπο να χρησιμοποιούν διάφορες κατασκευές ο τρόπος με τον οποίο μπορούν οι εφορίες να το αντιμετωπίσουν αυτό είναι να έχουν ακριβώς τις πληροφορίες για το τι συμβαίνει και τι γίνεται πού για να μπορούν να αντιμετωπίσουν με βάση τον εχώριο νόμο τους την κατάσταση. Η συνεργασία του Γκένσι είναι δεδομένη. Έχουμε υπογράψει πάρα πολλές διμερείς συμφωνίες ανταλλαγής πληροφοριών και αυτό είναι το ένα σκέλος, αλλά το άλλο σκέλος που είναι πολύ πιο πρόσφατο έτσι ως ε, επινόηση είναι η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών που άρχισε με την ε, αντίστοιχη οδηγία ε, και έχει φτάσει τώρα στις κοινέ προδιαγραφές για την κοινή δήλωση. Δηλαδή οι χώρες δεν θα πρέπει να μαθαίνουν εκ των προτέρων για τη φόρο αποφυγή και τη φόρο διαφυγή πριν ζητήσουν από εμά πληροφορίες. Εμείς θα τους στέλνουμε αυτόματα την πληροφόρηση σύμφωνα με το νέο σύστημα για το ποιες εταιρείε και ποια χαρτοφυλάκια και ποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εδρεύουν στο Γκένζε και στο Τζέρζι για να μπορούν να ελέγχουν τις υποθέσεις των φορολογουμένων και των πολιτών τους για να διαπιστώνουν αν υπάρχει φόρο διαφυγή ή φόρο Νομίζω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπο που μπορούμε να συνεργαζόμαστε με άλλα κράτη και δικαιοδοσίε. Τώρα, λέτε ότι δεν απαντήσαμε ουσιαστικά. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε ε, funds, συλλογικά συστήματα επενδύσεων. 2.000 άνθρωποι ασχολούνται με ένα πολύ μεγάλο βαθμό τέτοιων ε, συστημάτων συλλογικών επενδύσεων, επενδυτικών ταμείων, ε, με πολύ μεγάλα στοιχεία ενεργητικού. 2.000 εργαζόμενοι. Είναι αρκετοί, είναι σημαντική επιχείρηση. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε κάποιες θηρίδες μόνο με κάποιες ωραίες ταμπέλες γυαλιστερές και από πίσω τίποτα. Δεν ισχύει αυτό. Αν έχετε τέτοια εικόνα για τον Γκέρνζεϊ, έχουμε κόσμο που ασχολείται πολύ σοβαρά με αυτά τα ε, πράγματα. Στον Γκέρνζεϊ έχουμε 18.500 εταιρείες. 18.500 εταιρείες εδρεύουν. δεν είναι εκατοντάδες χιλιάδες όπως κυκλοφορεί, υπάρχει τέτοια αντίληψη. Ε, υπάρχουν αλλού τέτοιες, εμείς 18.500 μόνο έχουμε. Αυτά. Ελπίζω να απαντώ τουλάχιστον εν μέρη στην ερώτησή σας. Ίσως ο κύριος Πάολ να απαντήσει για τον Τζέρσι. Πολύ σύντομα. Όσον αφορά τις τραπεζικές καταθέσεις, νομίζω ότι όπως και σε άλλες καταστάσεις ε, οικοδομείται ένα επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης ε, που κάνει κάποιον ελκυστικό στην αγορά. Υπάρχουν πολλοί που ζητούν ένα ασφαλές καταφύγιο για τα χρήματά τους. Νομίζω όμως ότι το πιο σημαντικό είναι, και το είπαμε αρκετές φορές σήμερα, ότι όπως ε, είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΣΑ και όπως ε, είπε και το G20 ε, δεν υπάρχει πια κάποια κρυψώνα. Δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς από τις απαιτήσεις διαφάνειας και οποιοδήποτε τοποθετεί τα περιουσιακά του στοιχεία στο Γκένσι ή στο Τζέρσι θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα κοινά πρότυπα υποβολής εκθέσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Σβέν Κίγκολτ. Καταρχάς, να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω που ήρθατε, διότι γνωρίζουμε ότι δυστυχώς ε, οι νήσοι Κέιμαν αρνήθηκαν ε, να έρθουν σήμερα και δεν απάντησαν στις ερωτήσεις μας. Σας ε, ευχαριστώ λοιπόν εσάς που ήρθατε. Κύριε Πρόεδρε, κάνω λάθος. Πρόεδρος, πράγματι. Πρόκειται όμως για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Και ήδη αύριο θα ξαναστείλω επιστολή στις αρχές ε, των νήσων Κέιμαν για να φροντίσω να προσέρθουν. Καλή τύχη κύριε Πρόεδρε. Ή θα στείλω εσάς εκεί. Ναι, αλλά τώρα αφαιρέσατε από το χρόνο ομιλίας μου. Φυσικά και οι δύο αυτές δικαιοδοσίες έχουν ε, πρόσβαση στις ε, ευρωπαϊκές, κεφαλαιακές και άλλες αγορές. Από την ε, ανταλλαγή απόψεων κατάλαβα ότι σε σύγκριση με άλλους είσαστε μια σχετικά διαφανής δικαιοδοσία, αλλά είναι βέβαια πιο εύκολο να είναι κανείς διαφανής τη στιγμή που δεν φορολογεί. Διότι εάν σε πολλές περιπτώσεις εφαρμόζεται μηδενικός φορολογικός συντελεστής, τότε είναι εύκολο να το διαφανείς. Ούτε χρειάζεται να έχετε αποφάσει tax ruling εάν ο συντελεστή είναι μηδενικό, διότι ακριβώ το νόημα των αποφάσεων αυτών είναι να παρακάμψει κανεί την υψηλή φορολογία σε χώρε όπω οι κάτω χώρε ή το Λουξεμβούργο. Θα ήθελα όμω να σα ρωτήσω, θεωρείτε ότι ε, αποτελεί πρακτική καλής γειτονίας το να πέσει κανείς κάτω από το 10, 12 ή 5% ε, που είναι ο ελάχιστος φορολογικός συντελεστής στην Ευρώπη και θεωρείτε ότι είναι ε, καλή πρακτική γειτόνων να τραβάτε προς τα κάτω τους φορολογικούς συντελεστές. Και επίσης έχουμε την οδηγία κατά της ε, νομιμοποίησης παράνομων εξόδων ε, και ε, απαιτείται να υπάρχει μητρό πραγματικής κυριότητας όχι μόνο προσβάσιμο από τις διοικήσεις αλλά και σε τρίτους με κάποιο θεμητό συμφέρον. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιλέξει να είναι τελείως ανοιχτό το μητρό αυτό. Μπορείτε να μας πείτε πιο συγκεκριμένα εάν δεσμεύεστε κι εσείς να δώσετε πρόσβαση στο κοινό, στο μητρό αυτό ή τουλάχιστον σε ενδιαφερόμενους. Και επίσης, ε, από ό,τι κατάλαβα, έχετε ανταλλαγές με, το Ηνωμένο, ε, με τις Ηνωμένε Πολιτείε και έχετε συμφωνήσει ε, πάνω σε κάποια, σε, κάποια θέματα. Λοιπόν, θα υπάρχει πλήρης ισοδυναμία ΦΑΤΚΑ και από ό,τι καταλαβαίνω η Εστονία και η Πολωνία ε, αφαίρεσαν τις δικές σας δικαιοδοσίες από ε, τον κατάλογο φορολογικών παραδείσων. Ε, τι δραστηριότητες lobbying κάνατε για να το πετύχετε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κ. Πάουελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως αναφέρθηκε, από ό,τι γνωρίζουμε δεν υπάρχει συμφωνία για κοινό φορολογικό συντελεστή. Και από τον ΟΣΑ και τους G20 και την Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώσαμε ότι η θέση είναι ότι είναι θέμα κρατών οι φορολογικοί συντελεστές. Κάθε χώρα αποφασίζει ανάλογα με τις ανάγκες της. Εμείς θεωρούμε ότι έχουμε κάποια βάση, δεν έχουμε συμφωνίες διπλή φορολόγηση, έχουμε και μηδενικό συντελεστή φορολογικό για να αποφύγουμε διπλή φορολόγηση. Και όπως καταστήσαμε σαφές, μπορεί να είναι αποτελεσματική αυτή η διαδικασία αν υπάρχει επαρκής διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών με όλες τις νομοθεσίες. Αυτή είναι η άποψή μας. Και γίνεται όλο και πιο ευρέως αποδεκτή ότι το κλειδί είναι η διαφάνεια. Πολλές χώρες έχουν μηδενικό φορολογικό συντελεστή, άλλες νομοθεσίες έχουν πολύ χαμηλό φορολογικό συντελεστή και θα πρέπει μέσω διαφανείας να είναι ανοιχτή η θέση όλων. Η άλλη ερώτηση για το ΦΑΤΚΑ. Θέλουμε να συμμορφωθούμε με τις αρχές για ανταλλαγή πληροφοριών και υποβολή ε, αυτών. Είναι κάτι καλό και θα πούν ότι είναι καλύτερη η ρύθμιση από ότι το ΦΑΤΚΑ. Κυρίω βλέποντα τα έγγραφα του ΟΣΑ θα το διαπιστώσει αυτό, που γίνονται συγκρίσει μεταξύ του κοινού των προτύπων για την κοινή υποβολή πληροφοριών και το ΦΑΤΚΑ. Το νέο σύστημα είναι κάπω καλύτερο από το ΦΑΤΚΑ. Οπότε όλα τα κράτη-μέλη θα δέχονται πληροφορίε σύμφωνα με το σύστημα υποβολή πληροφοριών, το CRS. Όλοι συμμετέχουμε και θα αρχίσει η ζωή πληροφοριών το 2017. συμμετέχουμε πλήρως. Τέλος, για τις δικαιοδοσίες που μας έβγαλαν από τη μαύρη λίστα. Το έκαναν διότι κατανόησαν το επιχείρημά μας. Ποια είναι η θέση μας όσον αφορά τη συνεργασία μας και όσον αφορά τις μαύρες λίστες που καταρτίζονται για μη συνεργασία Βλέποντας ότι συνεργαζόμεθα εκτενώς, όπως και με την παρουσία μας εδώ, δεν υπάρχει λόγος να παραμείνουμε σε αυτές τις μαύρες λίστες. Συγγνώμη, δεν απαντήσετε όσον αφορά το Μητρό για την πραγματική διοκτησία. Α, ναι. Νομίζω ότι το ανέφερα κροθυγός προηγουμένως. θέλουμε να συμμορφωθούμε τη διεθνή πρακτική. Είδαμε την τέταρτη οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος και είδαμε τι αναφέρει. θα παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον τη δράση των κρατών μελών εν τη εφαρμογή της τέταρτης οδηγίας για το ξέπνο χρήματος. Και σύμφωνα με την αρχή μας περιπολιτικής καλής γειτονίας θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο με αυτό που κάνουν τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είμαστε ανοιχτοί σε αυτή τη φάση, διότι επί του παρόντος δεν ξέρουμε τι θα κάνουν τα ίδια τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εφαρμόζουν την οδηγία. Πρόεδρος. Τη κυρία Γκίγκολτ, για το Μητρό. Θα δημιουργηθεί τέτοιο Μητρό όπως απαιτείται. Τρίτα μέρη θα έχουν πρόσβαση στο Μητρό. Όχι μόνο δικήσεις. και για το Ηνωμένο Βασίλειο. είπατε, εξετάσατε την περίπτωση. Πέρασε πάνω από ένα χρόνο μετά τη συμφωνία. Θα έπρεπε να είχατε αποφασίσει αν θέλετε να είστε καλό γείτον σχετικά με αυτό ή όχι. Και αισθάνομαι ότι η απάντησή σα δεν είναι αρκετά σαφή. Απάντηση. Όσον αφορά την αφορά σε τρίτα μέρη, νομίζω ότι απάντησα στην ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Αλλά για μία ακόμη φορά. Η θέση μα είναι η εξή. Παρακολουθούμε την πορεία τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω σχετικά με την τέταρτη οδηγία περί ξεπλήματο χρήματο. Όπως καταλαβαίνουμε επί του παρόντο, δεν υπάρχει απέτηση σύμφωνα με την οδηγία για το κεντρικό μητρό αυτό που ήδη έχουμε και είχαμε ψηρά ετών να είναι δημοσία φύσεως, να είναι ανοιχτό. Τελούμε εν αναμονή των εξελίξεων. Τώρα όσον αφορά τα άλλα στοιχεία για τα ενδιαφερόμενα μέρη και την πρόσβασή τους θα παρακολουθήσουμε τι θα κάνουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πώς θα θεσπίσουν την νομοθεσία τους και αν ευθέτω χρόνο θα τοποθετηθούμε. Είμαστε ανοιχτοί. Θεωρούμε ότι ως καλούς γείτον πρέπει να ακολουθούμε το γείτονά μας. Άρα ε, ελπίζω να εννοείται το Ηνωμένο Βασίλειο. Απάντηση. Την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν και άλλοι γείτονε, λέει ο Πρόεδρο. Όχι μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο, έχετε και άλλους γείτονες. Τίμπο Ζάνη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απλοποιήσω όσο γίνεται τις ερωτήσεις μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο που ήρθατε σήμερα εδώ στην Επιτροπή μας και για τις προφορίες που μας δώσατε. Θα ήθελα να πω σε όλους ότι εγώ εκπροσωπώ ε, τους ε, Ευρωπαίους πολίτες και τους συμπατριώτες μου. Και ε, ο κόσμος θέλει να τα ακούει αυτά με τρόπο απλοποιημένο. Πρώτον λοιπόν, σύμφωνα με τη δική σας αντίληψη, ποιος είναι ένας ειλικρινής λόγος, η φιλοσοφία σας, η μεγάλη ιδέα, πώς το σκεφτήκατε, εν πάση περιπτώσει, να έχετε ένα τέτοιο μηδενικό φορολογικό συντελεστή για τις επιχειρήσεις. Τι σας ενέπνευσε γι' αυτό. Δεύτερη ερώτηση. Πάλι απλή. Είπατε ότι έχει, υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση για σας στην εσωτερική αγορά. Ωραία. Είστε πρόθυμοι να διαπραγματευτείτε ένα δίκαιο μερίδιο στον προϋπολογισμό της ενιαίας αγοράς όπως το κάνει για παράδειγμα η Νορβηγία. Συμμετοχή σας δηλαδή. Ευχαριστώ κύριε Σκρέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ποια είναι η φιλοσοφία ε, πίσω από το μηδενικό φορολογικό συντελεστή. Όπως είπε προηγουμένως ο κύριος ε, Πάουελ στην εισαγωγή του, τα νησιά είναι ε, ένας χώρος εισόδου κεφαλαίων στην Ευρώπη. Είναι ένα είδος αποθήκης, ας πούμε, κεφαλαίων και δεν θέλουμε να επιβάλλουμε διπλή φορολογία ε, στην επενδυτική δραστηριότητα. Διότι το Γκένζε και το Τζέρζι έχουν μια σχετικά περιορισμένη ε, ε, συμφωνία, αριθμό συμφωνιών για την διπλή φορολόγηση και ακόμα λιγότερο με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πιθανό σε περίπτωση που επιβάλαμε φορολόγηση σε συναλλαγές που διέρχονται από τα νησιά μας να μας εγκατέλειπαν. Ε, γιατί δεν θα υπήρχε αυτό ε, σε άλλες ε, δικαιοδοσίες και θα υπήρχε διπλή φορολογία. Ακριβώς λοιπόν, για να μην επιβάλλουμε και τους δικούς μας φόρους σε τέτοιου είδους συναλλαγές, επιτρέψαμε να φορολογούνται εκεί που εκτελούνται ή ασκούνται οι δραστηριότητες ή εκεί που ε, αποκομίζουν κέρδη οι εταιρείε έχει εισόδημα ο ε, πραγματικός δικαιούχος. Δεν θέλαμε δηλαδή να προσθέσουμε άλλο ένα στρώμα φορολογίας στη συναλλαγή. Όπως σας είπα, το έχω πει επανειλημμένα, αυτό δεν είναι ένα θέμα που αφορά τη δικαιοδοσία. Ε, στο βαθμό που ο καθένας έχει τις προφορίες, κανονίζει την πορεία του. Καταλαβαίνουν τι συμβαίνει, ποιος είναι ε, ο πραγματικός δικαιούχος και ποιος ε, αποκομίζει εισόδημα από αυτές τις συναλλαγές. Α, σε ό,τι αφορά τώρα την ενδεχόμενη ε, συμμετοχή μας στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μα δεν είμαστε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν νομίζω ότι είναι θέμα κάτι τέτοιο. Je Σας ευχαριστώ. Δεν είστε ούτε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, του ΕΟΧ. Οπότε δεν συντρέχει λόγος αυτή τη στιγμή για σας. Βεβαίως αν θέλετε μπορείτε να διαπραγματευτείτε κάτι διαφορετικό. Η Άννα και πάλι. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Μπορείτε να μας πείτε πώς είναι οι εφοριακοί που εργάζονται ε, στην επικράτειά σας. Εσείς παίρνετε αυτές τις αποφάσεις για αυτούς τους λεφτάδες εκεί ε, που έχουν κάποιες ε, ευνοϊκές ρυθμίσεις για ε, το, τη φορολογία των φυσικών προσώπων για το φόρο εισοδήματος. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Εσείς λέτε ότι είστε χρηματοπιστωτικά κέντρα και πραγματικά από αυτό ζείτε ως οικονομία στα νησιά σας. Αλλά πώς μπορείτε να είστε τόσο ε, απρόθυμοι να αλλάξετε κάποια πράγματα που πρέπει να αλλάξουν για να είναι αξιόπιστα τα χρηματοπιστωτικά κέντρα, ας πούμε σε ό,τι αφορά τη δημοσιοποίηση των πραγματικών δικαιούχων, των ιδρυμάτων και των καταπιστευμάτων. Γιατί πιστεύετε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η πιο απρόθυμη χώρα ε, που ε, ήθελε να μπει το θέμα των καταπιστευμάτων στην πρώτη οδηγία για την καταπολέμηση του ξεκλήματος ε, του χρήματος και το μητρό. Και επίσης, επιμένω στην προηγούμενη ερώτησή μου για τα ιδρύματα. Κάτω από ποιες συνθήκες, δηλαδή ποιες είναι οι απαιτήσεις για να ε, καταχωριστεί ένα ίδρυμα ή ένα φαντ. Ένα καταπίστευμα πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό, στόχο, δηλαδή πώς, πώς ιδρύει κάποιος ένα τέτοιο ίδρυμα. Είναι απλώς ένας φορέας, ένας ε, κατασκεύασμα για να φοροαποφεύγουν ή να φοροδιαφεύγουν ή ακόμα και να αποκρύπτουν εισόδημα, συγκεκριμένα την πηγή του εισοδήματος. Ευχαριστώ. Α, ξέχασα κάτι λέει η κυρία Γκόμας σκοπεύετε να συγκεντρώσετε και να, δημοσιοποιήσετε, να δημοσιεύσετε ε, στοιχεία, για στοιχεία ενεργητικού offshore ε, με βάση τη χώρα. Ας πούμε, εγώ θέλω να μάθω πόσοι Πορτογάλοι έχουν λογαριασμό ε, στα νησιά σας. Για να δούμε τι γίνεται εκεί. Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ονόματα θέλετε, λέει ο Πρόεδρος, ε. ε Κύριε Γκρέι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε σε ό,τι αφορά την εφορία ενδιαφέρουν και σε μέγεθος. Να σας εξηγήσω στον Κένζη τι γίνεται. Νομίζω απαντά επαρκώς. Η εφορία μας μία είναι. Και έχουμε περίπου 100 εφοριακούς που εργάζονται ε, ε, πλήρους και μερικής απασχόλησης. Και αυτός που είναι τελικά υπεύθυνος ε, για την διαχείριση της εφορίας είναι ο διευθυντή Φορολογίας Εισοδήματος που ήμουν εγώ μέχρι τα τέλη του 2015. Πραγματικά εγώ αποφάσιζα ε, για τα φυσικά πρόσωπα ε, και ποιο είχε ε, τη δυνατότητα φορολογικής ελάφρυνση ή φοροαπαλλαγής. Πραγματικά εγώ το αποφάσιζα αυτό σε ό,τι αφορά τα φυσικά πρόσωπα τώρα. Για τους πραγματικούς δικαιούχους των καταπιστευμάτων Κοιτάξτε, το καταπίστευμα δεν είναι από μόνο του ε, οντότητα. Είναι μια νομική ε, συμφωνία ε, και δεν έχει πραγματικούς δικαιούχους. Εκεί συμμετέχουν διάφοροι που συνεργάζονται και ελέγχουν στοιχεία ενεργητικού στο όνομα των δικαιούχων που τους έχουν εμπιστευτεί. Γι' αυτό είναι και καταπίστευμα και λέγονται trustees αυτοί και trust. Υπάρχει μια παρεξήγηση ευρέως διαδεδομένη που νομίζω στην οποία δεν αναφερθήκαμε και ίσως είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή να γίνει αυτό. Ο κόσμος συχνά μιλά για τα trusts ε, του Guernsey και του Jersey και τι εννοούν στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ένα trust το οποίο ε, εγγράφεται ε, στο δίκαιο του Γκένσε και Τζέρσι, δηλαδή χρησιμοποιώ τις δικαιοδοσίες ως παράδειγμα. Αυτό τι σημαίνει όμως. Αν υπάρξει καμιά διένεξη σε σχέση με το Trust, ε, για να λυθεί αυτό θα γίνει στα δικαστήρια του Γκένζη, γιατί υπάγεται στη δική μας δικαιοδοσία και στο δικό μας νόμο. Γιατί εκεί δικάζονται τέτοια θέματα και διεκπαιρεώνονται. Όντω, θα μπορούσατε, ας πούμε, να έχετε κάποιον που ζει στην άλλη άκρη του κόσμου, που δημιουργεί ένα τραστ, ε, το βάζει στο δίκαιο του Γκένζη και οι αρχέ Γκένζι μπορεί να μην έχουν ιδέα ποτέ για αυτό το τραστ. Μπορεί να μην έχει στοιχεία ενεργητικού, ε, ούτε η έδρα, ούτε οι ε, διαχειριστέ και ούτε κανένα από του δικαιούχου. Απλώ να είναι γεγραμμένο στο δικό μα δίκαιο και εμεί να αγνοούμε πλήρω την ύπαρξή του. Και αυτή είναι η δυσκολία να δημιουργήσει ένα μητρό των καταπιστευμάτων του Γκένζι, γιατί είναι πολλά τα οποία μα διαφεύγουν και δεν έχουμε καμία απολύτως ιδέα γι' αυτά. The, the issue of... Σε ό,τι αφορά ε, το θέμα των λεπτομεριών που δημοσιοποιούμε, δημοσιεύουμε ή τα δίνουμε στα κράτη-μέλη για τα τράσεις. Μα το κάνουμε αυτό. Από του χρόνου θα αρχίσει αυτό να γίνεται. Οι θεσμοί μας θα αναφέρουν ε, στην εφορία του Γκένζι και του Τζέρσι τις λεπτομέρειες σχετικά με το εισόδημα και τα στοιχεία ενεργητικού επενδυτών σύμφωνα με τους ε, κανόνες του Common Reporting Standard και στη συνέχεια αυτά θα διαβιβάζονται στι αρμόδιε φορολογικέ αρχέ των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και όλε τι άλλε δικαιοδοσίε με τι οποίε έχουμε συνάψει συμφωνία για ε, το σύστημα κοινή αναφορά. Έτσι, εν ευθέτω χρόνο όλα αυτά θα ε, είναι στη διάθεση των εφοριών των κρατών μελών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να απαντήσω για τα ιδρύματα σε ό,τι αφορά τα νησιά μας. Τα ιδρύματα καλύπτονται από την νομοθεσία και υπόκεινται σε γενική εποπτεία και ε, επισκόπηση. Ε, εμείς ε, τι είπαμε. Τον Ιούνιο του 2014 ήδη ο Πρωθυπουργός του Τζέρζι έκανε μια δήλωση για τα νησιά και είπε ότι δεν θέλουν ούτε χρειάζονται να καλύπτουν εκείνους που προχωρούν σε φοροδιαφυγή ή υπερβολική φοροαποφυγή. Τρία είναι τα στοιχεία αυτά και καλύπτονται και τα ιδρύματα. Ε, το βιομηχανικό επιμελητήριο έχει εκδώσει ένα κώδικα συμπεριφοράς και η ρυθμιστική αρχή και ένας από τους στόχους είναι να εντοπίσουμε πού οι δραστηριότητες αυτές ε, ε, μπορεί να είναι επιζήμιες για την φήμη και το κύρος της νήσου και τελικά η ίδια η κυβέρνηση ελέγχει ποιος δραστηριοποιείται γιατί ε, υπάρχουν και άδειες ε, εργασίας και άδειες ε, παραμονής. Και πραγματικά υπάρχει έλεγχος για το ποιος κάνει ποια δραστηριότητα και ποιος εγκαθίσταται και όλα αυτά ελέγχονται με βάση τα θεμητά συμφέροντα του νησιού και τη μελλοντική της φήμη και την ιστεροφημία της. Και έχουμε μια ολόκληρη δραστηριότητα, ένα ολόκληρο φάσμα ε, τέτοιων εμπορικών δραστηριοτήτων. Ο κύριος Λούκε, αντιπρόεδρος. Um, Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ο κύριος Πάουελ τόνισε και νομίζω ότι είχατε απολύτως δίκιο ότι είναι κυρίαρχο δικαίωμα κάθε χώρα να αποφασίζει ε, για τους φορολογικούς συντελεστές της. Μάλιστα. Και η δική μας δουλειά εδώ στην Επιτροπή δεν είναι τόσο πολύ να κοιτάμε το φορολογικό ανταγωνισμό, αλλά τα προβλήματα των κρατικών ενισχύσεων, που θα ήταν παράνομες, σύμφωνα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραία. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα τώρα είναι το εξής. Αυτά που συμβαίνουν στο Γκένζε και το Τζέρσεϊ μπορούν να θεωρηθούν κρατικές ενισχύσεις που μπορεί να μην είναι παράνομες με βάση τη δική σας νομοθεσία, αλλά σε εμά είναι παράνομες. Και εξ όσων είπατε εσείς κύριε Γκρέι, είπατε ότι υπάρχει πραγματική δραστηριότητα και το κατανοώ και εταιρείε που εδρεύουν εκεί δεν είναι απλώς μια θηρίδα ή μια, ε, μια ταμπέλα, αλλά είναι ουσιαστική εμπορική χρηματοπιστωτική δραστηριότητα. Η επιβολή όμως φόρου στους πολίτες και στις επιχειρήσεις τι σημαίνει ότι ε, ε, πληρώνεις φόρο για να χρησιμοποιείς τις δημόσιες υποδομές, δημόσιες υπηρεσίες ε, το δημόσιο, τα δικαστήρια κτλ. Αν έχετε λοιπόν πραγματικές δραστηριότητες των εταιριών σας γιατί δεν τις φορολογείτε. Εάν υπάρχει πραγματική δραστηριότητα και χρησιμοποιούν τις υποδομές σας αν υποθέσουμε ότι σημαίνει κάτι τέτοιο τις δημόσιες υπηρεσίες γιατί δεν τις φορολογείτε, γιατί δεν τους επιβάλλεται ένα φόρο για τη χρήση αυτών των υπηρεσιών. Και αν είναι ε, μηδενικός ο φορολογικός συντελεστής όταν χρησιμοποιούν τις υποδομές σας, δεν είναι κρυφές κρατικές ενισχύσεις αυτές. Ευχαριστώ, ο κύριος Γκρέι. Ευχαριστώ. Να σας δώσω λίγο το υπόβαθρο. Στο Γκένς είναι πάνω από 6.800 εργαζόμενοι στο χρηματοπιστωτικό τομέα, με την ευρεία του έννοια και με κάθε είδος δραστηριότητας. Ε, λιγότεροι από 1.900 εργάζονται στα τραπεζικά, 1.700 στα τραστ και στη διαχείριση και των επιχειρήσεων και όπως σας είπα προηγουμένως 2.000 στη διαχείριση των funds, των επενδυτικών ταμείων. Και επιπλέον έχουμε 700 που, χρησιμοποιούν, που εργοδοτούνται μάλλον ε, στις νομικές εταιρείες και 500 λογιστές. Δηλαδή έχουμε αρκετούς οι οποίοι εργάζονται ε, σε μόνιμη βάση και σε πλήρη απασχόληση. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λαμβάνουν μισθούς και ε, έχουν φορολογία φυσικών προσώπων, φόρο εισοδήματο. Και η πλειονότητα των φόρων μας προέρχεται από φυσικά πρόσωπα και ένα μεγάλο ποσοστό εκείνων από τους υπαλλήλους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εταιρείε και πώς εργάζονται και εργοδοτούν κόσμο, απασχολούν και εκείνοι ε, καταναλώνουν υπηρεσίες, άρα εμείς φορολογούμε το κάθε φυσικό πρόσωπο που κάνει χρήση κάποιων υπηρεσιών. Επίσης, ε, επιβάλλουμε ένα θετικό φορολογικό συνδελεστή σε κάποιες εταιρείες, 10% ας πούμε για τις τράπεζες. Ορισμένες ασφάλειες, ε, ορισμένες ε, χρηματοπιστωτικές ε, καταπιστεύματα και ορισμένα funds. Υπάρχει λοιπόν μια ολόκληρη δραστηριότητα στο χρηματοπιστωτικό τομέα που έχει φόρο 10%. Γενικά αυτές είναι περισσότερες επιχειρήσεις και που έχουν μόνιμη έδρα στο νησί και κάποιες από εκείνες που σας ανέφερα προηγουμένως με ουσιαστική δραστηριότητα. Υπάρχουν και κάποιες εταιρείες στην που ε, είναι κατοχής ε, ατόμων που δεν διαμένουν εκεί και έχουν δραστηριότητες τελείως εκτός της νήσου. Και αυτές έχουν να κάνουν με δραστηριότητες που υπόκεινται στο μηδενικό φορολογικό συντελεστή. Τώρα, αν θεωρείται αυτοκρατική ενίσχυση, όπως πολύ σωστά ρωτήσατε, και αναφέρατε στα σχόλιά σας, κρατικές ενισχύσεις είναι μια έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς δεν είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω ή να κρίνω αν κάτι τέτοιο είναι κρατική ενίσχυση. Είναι άγνωστος αυτός ο όρος και η έννοια στη δική μας νομοθεσία. Συμπληρωματική ερώτηση και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντηση. Θα ήθελα παρακαλώ να μου πείτε, αν σας κατάλαβα σωστά, είπατε ότι φορολογείται τα φυσικά πρόσωπα, εκείνους που εργάζονται στις εταιρείες, στη χρηματοπιστωτικό τομέα κτλ. Ωραία όλα αυτά. Και εκείνοι πληρώνουν για τις υποδομές και φορολογείται τα φυσικά πρόσωπα. Αλλά ένα φυσικό πρόσωπο που έχει εισόδημα από απόδοση κεφαλαίου χωρίς καμιά δραστηριότητα. Θα πληρώσει τον ίδιο φόρο για το ίδιο εισόδημα ενώ είναι ραντιέρης και δεν έχει χρησιμοποιήσει αυτή την, ε, ε, τις υποδομές, θα πληρώσει τον ίδιο φόρο με κάποιον που δουλεύει στην εταιρεία που εδρεύει στον Γκένσε. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το αντιλαμβάνεται η Ένωση αυτό, αυτό θεωρείται κρατική ενίσχυση. Και μια επιπλέον ερώτηση ο Πρόεδρος, αν ε, μου επιτρέπετε. Όταν λέτε ότι κάποιες εταιρείες έχουν φορολογικό συντελεστή 10%. Η φορολογική βάση ποια είναι, είναι εταιρική φορολογική βάση ή κάτι άλλο. Και έχετε μια αναφορά του Ηνωμένου Βασιλείου ή έχετε δική σας, έχετε δανειστεί από κάπου. Το δεύτερο να απαντήσω πρώτα γιατί μπορεί να βοηθήσει για να καταλάβουμε πώς έχει η κατάσταση. Οι εταιρείε και ε, τα πρόσωπα στο Γκέζε που εδρεύουν εκεί και οι εταιρείε μπορεί να είναι όμιλος που εδρεύει εκεί ή που είναι ιδιοκτήτης κάποιος κάτοικος Γκένζη, ε, φορολογούμε το εισόδημα. Δεν έχουμε φορολόγηση κεφαλαίου, ούτε ΦΠΑ έχουμε, ούτε τίποτα, ούτε φόρο του πλούτου, τίποτα. Μόνο φορολογία εισοδήματο έχουμε. Άρα η που ειναι ιδιοκτητη καποιο κατοικο γκενζη φορολογουμε το εισοδημα δεν εχουμε φορολογηση κεφαλαιου ουτε φπα εχουμε βάση για μια εταιρεία, είτε είναι στο 0%, το 10% και το 20%, είναι το παγκόσμιο εισόδημα της εταιρείας. Μόνο εισόδημα φορολογούμε και τίποτα άλλο. Ε, και έχουμε ε, απαλλαγές για πραγματικά έξοδα και για φορολογικά έξοδα, ας πούμε όταν υπάρχει υποτίμηση. Ε, πάντως δεν έχουμε τίποτα ε, που να δικαιολογεί ή να μπορεί να αφαιρέσει από το φόρο της μια εταιρεία κάτι που να είναι έκτακτη δραστηριότητα ή ασυνήθιστη. Και έρχομαι στη δεύτερη τώρα ερώτησή σας. Και το συνδέω με την προηγούμενη. Η κυβέρνηση του Γκιάνς έχει την εξή άποψη ότι το μεγαλύτερο του που έχουμε ε, στο νησί είναι οι εργαζόμενοι. Και οι περισσότεροι φόροι προέρχονται από φυσικά πρόσωπα και όχι από εταιρείε. Αν αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση το θεωρεί κρατική ενίσχυση, ε, τι να κάνουμε, θεωρήστε το. Ναι, αλλά με τη χρήση των υποδομών Α, είπατε ότι δεν έχετε υποδομές, αλλά δεν χρειάζεται να φορολογήσετε την ε, χρήση τους. Έχουμε υποδομές, πώς δεν έχουμε. Αλλά η κυβέρνηση επιλέγει να συλλέγει φόρους φορολογώντας φυσικά πρόσωπα το εισόδημά τους και ορισμένες εταιρείες. Πολύ σύντομα, επιτρέψτε μου. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω αυτό που είπε ο συνάδελφος. Στο Τζέρσι απασχολούνται 13.000 ε, στον χρηματοοικονομικό τομέα, περίπου 4.000 άτομα στις τράπεζες, 2.400 ε, σε νομικές υπηρεσίες ε, και 1.100 σε λογιστικές εταιρείες. Αλλά πρόκειται για περισσότερους, διότι λόγω της λόγω του ότι έχουμε ισχυρό χρηματοπιστωτικό τομέα, πολλοί άνθρωποι στο νησί στηρίζουν ακριβώς τον τομέα αυτών και παρέχουν υπηρεσίες προς τους ανθρώπους που εργάζονται στον τομέα αυτών και πρόκειται για άτομα που ζουν στο νησί και που πληρώνουν φόρο 20%. Αυτοί λοιπόν χρησιμοποιούν και στηρίζουν τις υποδομές. Και όπως ανέφερα νωρίτερα, το μερίδιο των εσόδων που ε, προέρχεται από εταιρικούς ε, φόρους ε, είναι σχεδόν ανάλογο του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο Τζέρσι η διαδικασία αυτή λειτουργεί πολύ καλά, διότι ως αποτέλεσμα έχουμε σχεδόν πλήρη απασχόληση και παρέχουμε καλές δυνατότητες απασχόλησης στους πολίτες, μας. Στους μας. Υπάρχουν επιχειρήσεις στο νησί, ε, που είναι η ιδιοκτησία μη κατοίκων ε, ε, χρησιμοποιούν τις υποδομές, υποβάλλονται σε φόρο ιδιοκτησίας και έτσι συνεισφέρουν στις υποδομές που χρησιμοποιούν, δρόμους κλπ. Ενώ οι επιχειρήσεις που είναι η ιδιοκτησία κατοίκων του νησιού και που για διανέμουν μερίσματα, ε, ε, πληρώνουν φόρους. Ε, δεν νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει ανισορροπία και δεδομένη στις δομή που έχουμε και της ισορροπίας που έχουμε βρει ανάμεσα στην εταιρική και στην προσωπική φορολογία. Νομίζω ότι όλοι συμβάλλουν στην υποδομή του νησιού. Ευχαριστώ. Αν δεν ζητά άλλο το λόγο. Α, η κυρία Γκόμες. Τα ιδρύματα λοιπόν και τα καταπιστεύματα φορολογούνται στα νησιά σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι μόνες οντότητες που φορολογούνται στο Τζέρσι είναι οι τα άτομα και οι επιχειρήσεις. Ενώ όσον αφορά τα καταπιστευματικά ταμεία, φορολογούνται ε, τα πρόσωπα πάλι και στις επιχειρήσεις και τα ιδρύματα φορολογούνται όπως οι επιχειρήσεις. Δηλαδή φορολογία 0% και όσον αφορά τους καταπιστευματοδόχους ε, αυτό εξαρτάται από τις πηγές εισοδήματος. Φορολογούμε ε, ε, σαν, οι δικαιούχοι να ε, το είχαν αυτό ως εισόδημα. Εξαρτάται λοιπόν από το εάν είναι κάτοικοι του νησιού οι δικαιούχοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα τις απαντήσεις που δώσατε και πρέπει να πω ότι έχω μπερδευτεί κάπως διότι φαίνεται σαν να ακολουθείτε όλους τους κανόνες διαφάνειας που είναι γνωστοί στην ανθρωπότητα, παρόλα αυτά όμως το Τζέρσι και το Γκέρνσι γενικά συνδέονται ε, με τη φοροαποφυγή και θεωρούνται φορολογική παράδειση. Μπορείτε να μου πείτε γιατί θεωρείτε ότι υπάρχει αυτή η παρανόηση ε, στους πολίτες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Πάουελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι η παρανόηση αυτή οφείλεται σε ιστορικούς λόγους. Αν πάμε πίσω στο χρόνο, θα διαπιστώσετε ότι σε σχέση με άλλες δικαιοδοσίες υπήρχε λιγότερη διαφάνεια, διότι δεν υπήρχαν διεθνή πρότυπα και υπήρχαν δραστηριότητε στο νησί που μπορεί να οδηγούσαν σε φοροαποφυγή ή επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Ε, τώρα λοιπόν, ε, όπως σας είπαμε σήμερα στις παρεμβάσεις μας ε, και όπως έχουμε απαντήσει και στις επιστολές μας, οι συνθήκες που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι αρκετά διαφορετικές. όπως υπόθηκε. Έχουμε υιοθετήσει τα στοιχεία διαφάνειας, έχουμε τα κοινά πρότυπα υποβολής εκθέσεων και θέλουμε να ακολουθήσουμε ε, την οδό αυτήν. Τώρα λοιπόν λέμε ότι ελπίζουμε ότι ήρθε η ώρα αυτή η ιδέα να μπει ε, κατά μέρο και να κοιτάξουμε το μέλλον. Εάν λοιπόν μας εξετάσετε υπό αυτό το πλαίσιο, δεν θα πρέπει να θεωρηθούμε φορολογικός παράδεισος. Άλλωστε, το, ο φορολογικός παράδεισος δεν, ε, δεν ε, αφορά μόνο τον φορολογικό συντελεστή. Ο φορολογικός παράδεισος είναι και ένα μέρος όπου μπορεί να κρυφτεί κανείς. Δεν θέλουμε λοιπόν να μας κατηγορήσουν ότι είμαστε μια κρυψώνα όσων θέλουν να φοροδιαφύγουν. Ευχαριστώ να ρωτήσω τον εισηγητή μας αν έχετε άλλες ερωτήσεις ή αν θέλετε να ε, ε, συνοψίσετε. Δύο πράγματα θέλω να θέσω. Νομίζω ήταν διεξοδική η συζήτηση, αλλά έχω δύο σημεία. Πρώτα απ' όλα για την πραγματική διοκτησία που συζητήσαμε ε, εκτενώς. Θα γνωρίζετε Φαντάζομαι ότι ο Ντέβιτ Κάμερον, ο Βρετανός Πρωθυπουργό το 2014 τον Απρίλιο είχε μεταβεί και είχε αναφερθεί στη σημασία που έχει ένα κεντρικό μητρό όσον αφορά την πραγματική διοκτησία και να υπάρχει και δημόσια πρόσβαση. Αυτό είχε πει στην επίσκεψή του. Αυτό αντιστοιχεί σε εσά. Και μετά τη σημερινή συζήτηση εκπλήσωμε που δεν έχει εφαρμοστεί αυτή η σύσταση που έκανε ο Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου. Και έστειλε επιστολή και λέει σε αυτή που σας απέστειλε ο Ντέιβιτ Κάμερον. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι πληροφορίες περί επιχειρήσεων και πραγματικών διοκτητών να διατίθεται δημοσία θα δώσει επιχειρήσεις και στους ανθρώπους ποιος πραγματικά είναι ιδιοκτήτης και ελέγχει την επιχείρηση. Και είναι πιο εύκολο για νομικούς, τράπεζες κλπ. να ε, μπορούν να ενημερώνουν σωστά τους Πελάτε του, Θα ρίξει φω σε εκείνου που έχουν παράσχει ψευδεί πληροφορίε και έτσι αντιμετωπιστεί το έγκλημα όταν αυτό συμβαίνει και θα αποτρέπονται οι άνθρωποι να δίδουν ψευδείς πληροφορίες. Θα μειωθεί το κόστος των ερευνών για τις αρχές της φορολογικής και επιβολής του νόμου και εδώ και σε άλλες χώρες, κυρίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, αν είναι πιο εύκολη η πρόσβαση στις πληροφορίες όταν διενεργείται μια έρευνα. Αυτό ήταν το επιχείρημα του Ηνωμένου Βασιλείου τότε το 2014. Αλλά δεν θέλετε, διστάζετε πάρα πολύ να δίνετε πληροφορίες από το Κεντρικό Μητρό περί πραγματικής ιδιοκτησίας. Γιατί, είναι η ερώτησή μου. Μετά αν δείτε τους αριθμούς, που είναι πάντα χρήσιμο κάτι τέτοιο. Το 2007, σύμφωνα με τον Colin Powell, οι, τα, τα διάφορα τα, οι τράπεζες, οι offshore και άλλοι φορείς είχαν περίπου 700 εκατομμύρια, 800 εκατομμύρια λίρες είναι περίπου ε, το μισό με την επιχειρηματική, με την οικονομική παραγωγή του Ηνωμένου Βασίλειου. Και αυτά, αυτά τα χρήματα βρισκόταν στο Τζέρσι. Με τόσο πολλά στοιχεία ενεργητικού σε καταπιστεύματα και σε τραπεζικά ιδρύματα Δεν θεωρείτε ότι αυτοί οι πόροι βρίσκονται εκεί για λόγου φορολογικού. Γιατί να έρθουν αυτοί οι φορεί εκεί. Γιατί να έχουν τόσο τεράστια ποσά εκεί, αν δεν ήταν ε, σκοπός σκοπό του η αποφυγή του φορού. Τεράστια ποσά. Πάρα πολύ μεγάλα ποσά βρίσκονται εκεί. Και γιατί έρχονται, αν όχι ε, για φορολογική διευκόλυνση. Ο καλός καιρός, λέει ο Πρόεδρος, των ίσων της μάχης, ο κ. Πάολ, για να απαντήσω στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο έθεσε σαφώς τη θέση του. Μετά την σύνοδο GH στο Λόκερεν. Προσπάθησαν να πείσουν τους G8 και μετά τους G20 και την Ευρωπαϊκή Ένωση φαντάζομαι ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν την πορεία τους για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων περί πραγματικής ιδιοκτησίας. Με την πάροδο του χρόνου όμως στη συζητήση με τον Αμένο Βασίλειο κατανόησαν ότι τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο καλά όσο θα ήλπιζαν και είναι παράλογο να περιμένουν να προχωρήσουμε εμείς και να ακολουθήσουμε την πορεία που ακολουθείται στον κόσμο. Το Ενωμένο Βασίλειο θα ήθελε να ευθέτω χρόνο να δημοσιοποιείται αυτά τα στοιχεία αλλά κατανόησαν ότι λόγω των περιστάσεων έπρεπε να ακολουθήσουμε σταδιακή προσέγγιση. Καταρχάς να δημιουργήσουμε κεντρικό μητρό και μετά ανάλογα με το αυτό που κάνουν οι άλλες χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσουμε προς δημόσια δημοσιοποίηση ε, των στοιχείων του μητρό. Και εμείς έχουμε ήδη το δημόσιο Μητρό αυτό, θα μπορούσαμε να συμμορφωθούμε, για τα 700 με 800 δις ε, λίρες και με το επιχείρημα ότι μάλλον για λόγους φορολογικούς ήρθαν τα χρήματα. Να σας πω γιατί δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Αν πάρτε τις αποταμιεύσεις των τραπεζών, σημαντικό ποσό. Οι πληροφορίες των τραπεζών θα διατεθούν στις ενδιαφερόμενες χώρες, οι υπήκοοι των οποίων έχουν καταθέσει τα χρήματά τους στο Τζέσσε και στο Γκένσε. Και πολύ συχνά για άλλους λόγους, όπως είναι η πολιτική σταθερότητα και τα τόκοι όσον αφορά τις καταθέσεις ίσως εκεί ε, να καλύπτεται τα θέματα τα φορολογικά. Και το Γκέντζι μαζί με άλλες χώρες και με πολλά κράτη-μέλη και με το Ηνωμένο Βασίλειο δεν φορολογεί τους τόκους που καταβάλλονται στους μη κατοίκους. Υπάρχει είναι ανοιχτή θέση μας όσον αφορά τις αποταμιεύσεις. Δεν καταδίδεται τα χρήματα για λόγους φορολογικούς, διότι όλα είναι πολύ διαφανή. Για τα καταπιστεύματα. Μεγάλο ποσοστό των χρημάτων αυτών. Έχουμε δημιουργήσει φήμη, τεχνογνωσίες, εμπειρίες όσον αφορά τη διαχείριση των καταπιστευμάτων. Σε μεγάλο βαθμό τα καταπιστεύματα αυτά φορούν τη διαχείριση πλούτου και προστασία αυτούς. Βασίζονται σε κεφάλαιο και όχι σε εισόδημα. Δεν, δεν υπόκεινται σε φορολόγηση κεφαλαίων. Διαθέτουν τις πληροφορίες σε άλλες χώρες. Και αυτά τα καταπιστεύματα δημιουργούνται από κάποιους που επιδιώκουν ασφάλεια και κυρίως φεύγουν από περιοχές με πολιτική αστάθεια. Και ο φόρος δεν είναι το βασικό κίνητρο για τη διαμόρφωση, για τη δημιουργία αυτών των καταπιστευμάτων. Σε συνέχεια αυτόν που είπε ο κύριος Πάουελ, ιστορικά θυμάμαι τότε που το Γκένσι είχε αρχίσει να διαπραγματεύεται συμφωνίες ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών το 2001 και αρκετοί τότε είπαν ότι αυτό θα σημάνει το τέλος του χρηματοπιστωτικού τομέα του Γκέρνση, διότι ε, βασίζεται αποκλειστικά στην ε, χαμηλή φορολόγηση. Αλλά αυτό δεν συνέβη. Και το 2005, κατά την αναθεώρηση της οδηγίας, ε, πολλοί είπαν ότι αυτό είναι το τέλος του Γκέρνση όσον αφορά τους πελάτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε συνέβη αυτό με τις 60 ε, συμφωνίες ε, ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών που ε, συνάψαμε ούτε τις συμφωνίες διπλής φορολογίας. Και αυτό συνάδει με αυτό που είπε ο κύριος Πάουελ, ότι το μεγαλύτερο μέρος της διαφάνειας συνδέεται με την φορολογία. Και τώρα προχωράμε και στα BEPS. Η θέση λοιπόν είναι ότι ο τομέας αυτός δεν στηρίζεται αποκλειστικά στη χαμηλή φορολογία όπως θέλουν να ισχυρίζονται οι επικριτές μας. Ευχαριστώ. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι. Δεν ζητά άλλο το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους δύο α, ομιλητές. Καταλαβαίνουμε καλύτερα την κατάσταση που κρατεί στο Τζένσι και στο Γκένζι. Είναι δύο μικρά νησάκια όπου η ιστορία και η γεωγραφία τα έθεσε σε κάπως ιδιαίτερη θέση και αρκετοί από τους συναδέλφους μας εξεπλάγησαν που δεν υπάρχει εταιρικός φόρος, corporate tax. Αλλά λόγω των αναγκών της νομοθεσίας σας, το income tax, ο φόρος εισοδήματος, αρκεί για τη χρηματοδότηση των δημοσίων υπηρεσιών σας. Ταυτόχρονα, και αυτό εξαρτάται από την κυριαρχία σας, θα πρέπει εμείς να φροντίσουμε το ώστε οι γειτονικέ νομοθεσίες Ευρωπαϊκής Ενώσης να μην επιτρέπουν σε επιχειρήσεις ανεξάρτητα της εθνικότητας τους που κάνουν κέρδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφεύγουν την καταβολή των φόρων όσον αφορά αυτά τα κέρδη. Αυτό είναι και το νόημα όλων των προσπαθειών μας. Μας όταν λέω εννοώ Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ΣΑ εδώ και αρκετά χρόνια και γνωρίζετε, αλλά σας το αναφέρω, όπως θα το έλεγα και στις προσωπικότητες που θα έρθουν αύριο εδώ, θα πρέπει να καταλάβετε ότι αλλάζει η εποχή, αλλάζουν οι εποχές και ότι η περίοδος κατά την οποία κάποιες χώρες μπορούσαν να προβούν σε φορολογικό ανταγωνισμό για να προσελκύσουν επιχειρήσεις ή προσωπικότητες ε, πλούσιες ήταν μια περίοδος που πια άλλαξε και από την πλευρά των εκλογέων μας, διότι όλοι ανήκουμε σε δημοκρατίες και εκπροσωπούμε τους πολίτες. Υπάρχει βούληση λοιπόν στους πολίτες για διαφάνεια και για δικαιοσύνη. Κατανοούμε απολύτως αυτά που είπαν και πολλοί που παρενέβησαν και την πρόεδρος Λούκε ότι κάθε χώρα είναι κύρια της φορολογίας της και των φορολογικών ε, συντελεστών που εφαρμόζει. Αντιθέτως, αυτό που δεν είναι πλέον αποδεκτό για τις ε, κυβερνήσεις είναι ότι κάποιες χώρες κλέβουν φορολογικό υλικό από το γείτονα το ΣΥΠΗΝ. Και για τους πολίτες βλέπουν ότι αυτή είναι μεγάλη αδικία. Υπάρχουν αυτοί που πληρώνουν, οι μικρές και μεσές επιχειρήσεις, σε σχέση με τις μεγάλες πολυεθνικές που καταφέρνουν να αποφύγουν τις πληρωμές. Λοιπόν, ε, θέλουμε να ανταποκριθούμε στα αιτήματα περί διαφανείας και δικαιοσύνης των συμπολιτών μας. Αυτό αληθεύει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ισχύει και το βλέπουμε μέσω των εργασιών του ΟΣΑ. Και υπάρχει πολιτική βούληση για να στηρίξουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προτάσεις που έκανε και συζητήσαμε εκτενώς σήμερα, τις έκανε αρχές του έτους όσον αφορά όσον αφορά το BEPS ε, Action Plan που πρέπει να ενσωματωθεί και να εφαρμοστεί μέσω εθνικών νομοθεσιών. Και κάτι που συστήσαμε εμείς στην αρχή. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει προτάσεις στο δεύτερο εξάμεινο, προτάσεις που αφορούν την εναρμόνιση της φορολογικής βάσης των φόρων επιχειρήσεων, του corporate tax εντός τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Θα διοργανωθεί λοιπόν μια συνάντηση για ανταλλαγή απόψεων με συμμετοχή εκπροσώπων των 28 Εθνικών Κοινοβουλίων με αυτό το θέμα. Θα λάβει χώρα στις 18 Απριλίου, σας το λέω για να σε ενημερώσω. Θα συμμετάσχουμε επίσης σε μια διακοινοβουλευτική συνάντηση επί του θέματος που διοργανώνει ο ΩΣΑ στις 2 Μαΐου εις Παρισίους. Εκεί όλες οι κυβερνήσεις, όλες οι χώρες που επεξεργάστηκαν το BEPS Action Plan θα προσκληθούν να συμμετάσχουν και κατά τη διάρκεια του Μαΐου θα μεταβούμε εις ΕΠΑ για να συναντήσουμε τις αρμόδιες επιτροπές ε, των δύο βουλών ε, του Capitol Hill για να συνεννοηθούμε για τις δράσεις μας για να δούμε πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν σε διεθνή κλίμακα αυτά τα θέματα. Επανειλημμένα εκφράσατε την θέλησή σας του Τζέρσε και του Γκένστρε, τη θέληση των χωρών, των νήσων αυτών να συμμορφωθούν και να συμμορφωθούν με τις ε, συστάσεις και είμαστε πεπισμένοι ότι όλοι μαζί θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην αλλαγή νοτροπίας και σε αυτή την ήσυχη μετάβαση. Σας ευχαριστώ. Ας μείνουμε σε επαφή, ας συνεχίσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών, αυτό σας προτείνω, όσον αφορά τις δράσεις που ακολουθούμε και η μεν και η δε. Σας ευχαριστώ. Ας λήξει εδώ η συνεδρίαση και θα τα ξαναπούμε αύριο στις 9 για την ακρόαση των τριών άλλων ε, δικαιοδοσιών. Λοιπόν, πέρα στη συνεδρία σας και καλό σας βράδυ.